Αγαπητοί συνάδελφοι, αν είστε έτοιμοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Παγκόσμια ημέρα, είδα το σήμερα. Ξεκινάμε με την στη διάταξη. Αλλά θα ήθελα καταρχάς για τους δανούς συναδέλφου, να πω ότι τα δανεικά δεν έχουν καμπίνα σήμερα. Είναι μόνο παθητική θα ακούτε μόνο, θα μπορείτε να μιλάτε μόνο. Θα μπορείτε μόνο να μιλάτε δανεικά, αλλά όχι να ακούτε διερμηνία. Α, η κυρία Ρώσπα, είναι ευχαριστημένος εκ του. Καλώς. Και πάω στο σημείο 18 και 19 μαζί. Ξεκινώντας με την κυρία Μακ Εύαν την εισηγήτριά μας. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν έχουμε πολύ μελή επιτροπή στην Ελλάδα, έχουμε μεγάλη προσέλευση. Το θέμα όμως που θα συζητήσουμε είναι άκρο σημαντικό. Και ίσως να αναρωτιούνται οι συνάδελφοι γιατί πάλι συζητούμε τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Ενώ είχαμε συμφωνήσει με το Συμβούλιο σε νέα νομοθεσία. Μόλις πριν από 18 μήνες. Ναι, είναι αυτοί που μιλάνε Είχαμε συμφωνήσει λοιπόν σε νέα νομοθεσία η οποία βελτιώνει τη, σημαντικά την ασφάλεια των φαρμάκων σε σχέση με το παρελθόν. Πλην όμως από τη δημοσίευση της ε, νέας νομοθεσίας θα θυμούνται οι συνάδελφοι. Προέκυψε μεγάλο σκάνδαλο στη Γαλλία, υπόθεση Mediator, και θα σας πω και λίγο περισσότερα πράγματα για την υπόθεση αυτή και γιατί είναι σημαντική για την ε, νομοθεσία μας, αλλά ε, μετά την υπόθεση αυτή στη Γαλλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια επαλήθευση μια ανάλυση της υπόθεσης, το λεγόμενο stress test και θα θυμάστε ότι είχαν έρθει οι εκπρόσωποι της Επιτροπής για να μας παρουσιάσουν τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης. Η Επιτροπή λέει ότι και τη, η νέα αυτή νομοθεσία έχει επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην, μακρο, στην φάρμακοεπαγρύπνηση, χρειάζονται ακόμη βελτιώσεις. Θα συμφωνήσω εγώ με την Επιτροπή λοιπόν σε αυτό. Υπάρχουν κάποιοι τομείς ίσονες ίσως, στους οποίους χρειάζεται να κλείσουμε κάποια ακόμη αναπομείναντα παραθυράκια. Από την υπόθεση με διατόρα αυτό που μάθαμε ήταν ότι η επιχείρηση αυτή, η εταιρεία αυτή, είχε αξιοποιήσει κάθε παραθυράκι, κάθε χαραμάδα στην νομοθεσία για να ε, προχωρήσει στη διάθεση των προϊόντων της. Και αυτό κάλυψε άλλωστε και η ανάλυση της υπόθεσης. Είχαμε συζητήσει το θέμα με τους κοιόδης συγκητές και είχαμε συμφωνήσει ότι θα μπορούσαμε χωρίς βραδιπορία να καταλήξουμε σε μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση και ή δυνατόν, ή δυνατόν σημαίνει εφόσον και το Συμβούλιο συνεργαστεί, μπορούμε να έχουμε έτοιμη την νομοθεσία για να τεθεί σε ισχύ από τον Ιούλιο ήδη εφέτος. Εφόσον όλοι συνεργαστούν λοιπόν για τι πρόσθετε αυτέ αλλαγέ στην νομοθεσία. Αυτή είναι και η δική μου πρόθεση, Πρόεδρε, αλλά πρέπει να είναι και σωστή η νομοθεσία αυτή. Φορά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε δηλαδή να παραμείνουν οι αδίποτε παραθυράκια. Τι είναι η υπόθεση Μεντιατός. Ένα αστείο ήταν τη γαλλική επιχείρηση Σερβιέ ε, ήταν ένα φάρμακο, ναι. της γαλλικής επιχείρησης Servier που είχε πάρει άδεια, ε, ήταν ένα φάρμακο για διαβήτη τύπου Β, κυκλοφορούσε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και Ήδη υπήρχαν κάποιες ενδείξεις από το 1988 ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανομαλίες, σε προβλήματα στην καρδιακή βαλβίδα. Συνέχισε όμως παρά αυτές τις ανησυχίες να κυκλοφορεί και να σταγογραφείται το φάρμακο αυτό και όχι μόνο για τους πάσχοντες από διαβήτη τύπου Β, αλλά και γενικότερα για όποιον ήθελε να ε, χάσει βάρος. Και έτσι το 2009 όταν ε, ουσιαστικά έγινε και η ενδελεχής εξέταση των διαφόρων ανησυχιών ε, των σχετικών με την ασφάλεια του φαρμάκου, απεσήρθη από την αγορά. Εν τω μεταξύ όμως 5 εκατομμύρια ανθρώπων είχαν υποστεί προβλήματα λόγω της χρήσης αυτού του φαρμάκου, το οποίο ήταν το πιο ευρέως συνταγογραφούμενο φάρμακο στην Ευρώπη. Ενώ υπήρχαν προβλήματα ήδη ενδείξεις σημαντικές και από τη δεκαετία του 90 πως ε, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην καρδιακή βαλβίδα και υπολογίζεται ο αριθμό των νεκρών μπορεί να είναι από 500 έως 2.000 λόγω της κρίσης αυτού διατόρ. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να επισημάνω ότι πολλές φορές μέσα στις ρυθμιστικές αρχές, στα θέματα φαρμάκων ε, μπορεί να εκφράζονται ανησυχίες για κάποιο φάρμακο. Οι ΗΠΑ, σε παραδείγμα, είχαν αποσύρει πολλά χρόνια πριν αντίστοιχο φάρμακο Πλην όμως στην Ευρώπη δεν λειτουργήσε έτσι το σύστημα. Και γιατί, διότι εάν ανατρέξουμε στις αρχές δεκαετίας του 2000, είχαμε ένα σύστημα επαγρύπνησης φαρμακοεπαγρύπνησης όχι επαρκώς αναπτυγμένο στην Ευρώπη και δεν υπήρχαν επαρκή μέσα για να ληφθεί δράση σε περίπτωση προβλήματος ε, προκαλούμενο από ένα φάρμακο. Το Mediator λοιπόν δεν είχε ζητηθεί επαρκώ. Είχε ζητηθεί σε έναν βαθμό στην Ισπανία το σύνολο των ανησυχιών που προξενούσε σε αυτό το φάρμακο και έτσι η εταιρεία Σερβιέ αποφάσισε μονομερό να το αποσύρει από την αγορά και να μην ξανακαταθέσει αίτηση για διοδότηση στην Ισπανία και την Ιταλία μετά το 2003. Άρα εξαφανίστηκε από την αγορά το 2003 το φάρμακο. Τα λοιπά κράτη-μέλη ενημερώθηκαν ότι απεσύρθη από την Ισπανία και την Ιταλία το φάρμακο την εποχή εκείνη Πλην όμω δεν έγινε και διερεύνηση των προβλημάτων σχετικών με την ασφάλεια του φαρμάκου αυτού, γιατί εκείνη την εποχή και με την νομοθεσία όπω ίσχυε, εάν αποφάσισε να αποσύρει μια εταιρεία ένα φάρμακο από την αγορά, δεν γινόταν τίποτα. Δεν υπήρχε ανάγκη δηλαδή για περαιτέρω μέτρα. Έλεγε ότι για εμπορικού λόγου αποσύρει το φάρμακο από την αγορά η εταιρεία και δεν γινόταν περαιτέρω διερεύνηση και ότι υπήρχαν στο παρελθόν ήδη είχαν γίνει συζητήσει για ανησυχίε και προβλήματα σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Ε, και μόνο το 2009, όταν κάποιος, κάποιοι Γάλλοι υπάλληλοι, κρατικοί υπάλληλοι στην Νότια Γαλλία άρχισαν να εξετάζουν πιο προσεκτικά το ζήτημα, προέκυψε η υπόθεση, απεσύρθη ουσιαστικά το φάρμακο και τώρα ανατρέχοντας στο παρελθόν Βλέπουμε τις συνέπειες με την, ε, με την παρέτηση του επικεφαλής της Γαλλικής Αρχής ε, Φαρμάκων, του Γαλλικού Φορέα Φαρμάκων και βλέπουμε πόσο μεγάλη καθυστέρηση ε, υπήρξε σε σχέση με το φάρμακο αυτό. Και για να επανέλθω στην νομοθεσία, επειδή υπήρχαν κάποιε ανησυχίε σχετικέ με την ασφάλεια του φαρμάκου στα τέλη τη δεκαετία του 90 και στι αρχέ τη δεκαετία του 2000, ζητήθηκε από την αρχή μια μελέτη από τη Mediator για τον Μεντιατόρ μάλλον. Δηλαδή μπορεί να τεθεί στην αγορά το φάρμακο και να ζητηθεί από την αρμόδια αρχή ε, επιπλέον μελέτη ασφάλειας του φαρμάκου. Ζητήθηκε λοιπόν η σχετική μελέτη το 2001. Αν δεν κάνω λάθος, κοιτάω στα χαρτιά μου. Το 2001 λοιπόν ζητήθηκε η μελέτη που θα έπρεπε να κρατήσει ένα χρόνο περίπου Το 2001 λοιπόν η Γαλλική, ο Γαλλικός Οργανισμός Φαρμάκων ζήτησε τη μελέτη για το Μεντιατόρ, αλλά η Γαλλική Γερουσία μας λέει ότι μόνο το 2006 ξεκίνησε πραγματικά αυτή η μελέτη. Και το 2009 ολοκληρώθηκε μόνο και παρουσιάστηκαν τα σχετικά αποτελέσματα. Ε, και τότε βέβαια αποσύρθηκε από την αγορά το φάρμακο. Επί 8 χρόνια λοιπόν ε, καθυστέρησε η ε, υπόθεση αυτή και μετά απεσύρθηκε το φάρμακο από την αγορά. Όταν λοιπόν πρώτο η πρόταση για τη φαρμακοεπαγρύπνηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, έλεγε η πρόταση ότι Εάν ένα φάρμακο υπαχθεί σε κάποια μελέτη, είτε στην αρχή, είτε στη διάρκεια της αθήσης στην αγορά, θα πρέπει να σημειωθεί με ένα μαύρο μάλιστα σύμβολο, με ένα μαύρο τρίγωνο, στον κατάλογο, τον ειδικό κατάλογο των φαρμάκων για τα οποία υπάρχουν ανησυχίε. Και έτσι γνωρίζει ο κόσμο, ο, ο καταναλωτή, ότι το φάρμακο αυτό έχει μεν λάβει άδεια, αλλά υπάρχουν ακόμη κάποια ζητήματα που θα πρέπει να επιληθούν. Στήριξε την Επιτροπή το Κοινοβούλιο στην πρόταση αυτή μας από την πρώτη ανάγνωση. Στις διαπραγματεύσεις όμω με το Συμβούλιο απερίφθη η σχετική διάταξη. Μία πρόταση λοιπόν που επαναφέρει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ακριβώς αυτή η επανασύνδεση του φαρμάκου, ε, στον, η επανεγραφή του φαρμάκου στον κατάλογο των υπόπτων προϊόντων και η επισήμανση ότι υπάρχει ανάγκη για μελέτη ασφάλειας. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό, διότι Εάν έχει το μαύρο τρίγωνο, το μαύρο αυτό σύμβολο το φάρμακο, γνωρίζει ο καταναλωτή ότι είναι καινούριο φάρμακο ή πρέπει να επανεξεταστεί και άρα και ο γιατρό ή όποιο αρμόδιο ε, από το υγειονομικό προσωπικό έχει την σχετική ευαισθητοποίηση και μπορεί να επισημάνει κάποιες παρενέργειες που ενδεχομένω παρατηρεί. Επιπλέον, είναι κίνητρο το μαύρο τρίγωνο για την εταιρεία, τη φαρμακοβιομηχανία δηλαδή, να επανεξετάσει και να ε, κινηθεί ταχύτερα, να μην περάσουν 8-9 χρόνια όπως έγινε τώρα, με συνέπειες βέβαια για την υγεία και την ασφάλεια των ε, πολιτών ε, για την περίπτωση του Μεδιατόρ και άλλωστε το επισημάνουν και οι Γάλλοι στη μελέτη τους. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η Επιτροπή με την νέα νομοθεσία, δηλαδή επαναφέρει την αρχική πρόταση για την υπαγωγή του φαρμάκου στον κατάλογο των εντατικά παρακολουθούμενων αυτών δηλαδή που έχουν ανάγκη για επιπλέον μελέτες ασφάλειας. Στην περίπτωση της Σερβία τι συνέβη. Η Σερβία δεν ξανά έκανε αίτηση για να πάρει και πάλι την άδεια διάθεση στην Ισπανία και την Ιταλία. Όταν το απέσυρε, όπω είπα, δεν έγινε τίποτα. Δεν προβλέπει διαδικασία καμία δυνατότητα για τι χώρε, τις λοιπές χώρες διάθεσης να πούνε γιατί το αποσύρατε από εκεί. Και άρα ε, αυτό αλλάζει τώρα και έχουμε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία κατεπήγοντο, όπου θα πρέπει να δοθούν εξηγήσει, αν υπάρχουν λόγοι ασφάλεια, μέσα από αυτή την κατεπίουσα διαδικασία η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων και ιδιαίτερα η ε, Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνασης και εδώ σημειώνω ότι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό ήταν το ότι ενισχύσαμε αυτή την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνασης γιατί δεν ήταν τόσο ισχυρή στο παρελθόν μέσα στην ε, υπηρεσία φαρμάκων. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι και έτσι εάν υπάρξουν διαπιστώσεις σχετικές με την ασφάλεια, με προβλήματα ασφάλειας, τότε συζητείτε αυτό σε επίπεδο ε, εμπειρογνωμόνων. Και βλέπουμε ότι πολλές φορές ζητήματα που συζητούνται μεταξύ των ειδικών πλέον με την πρόταση αυτή βγαίνουν και συζητούνται ουσιαστικά στην Τράπεζα των Συζητήσεων. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίπτωση Σέρβια, Σερβία ήταν ότι η, στη συγκεκριμένη περίπτωση η εταιρεία είπε ότι δεν ε, επανακατέθεσε αίτηση για άδεια διάθεση στην αγορά στην Ισπανία και την Ιταλία για λόγους εμπορικούς για λόγους marketing. Αλλά τώρα αυτό το θέμα αμφισβητείται βέβαια και είναι αντικείμενο τη συζήτησης, ε, τη όλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει στη Γαλλία. Μάλλον δεν ήταν αυτό, ήταν για να αποφύγει τι σχετικέ διαδικασίε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θα θέλω να επισημάνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα έπρεπε, θα πρέπει, οτιδήποτε τώρα γίνει με τη νέα νομοθεσία, όταν μια εταιρεία αποφασίσει να μην καταθέσει και πάλι αίτηση για διάθεση στην αγορά ενό προϊόντο, να εξηγεί και γιατί. Και μάλιστα ρητά να καλείται να δηλώσει, εάν δεν πρόκειται για λόγους ασφαλεία, ότι δεν πρόκειται για λόγους ασφαλείας. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τις προτάσεις της τώρα και νομίζω ότι είναι σωστές, είναι εύλογες προτάσεις. Δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα παραθυράκι, κανένα, καμιά χαραμάδα στην νομοθεσία και τούτου. Θα κοιτάξουμε με πολύ μεγάλη προσοχή τη διατύπωση. Από πλευρά στο Συμβούλιο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι πολύ επιφυλακτικό προς το ζήτημα του μαύρου συμβόλου, του μαύρου τριγώνου. αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα και πάλι με το Συμβούλιο όταν έρθει η ώρα του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί εγώ θα ζητήσω από το Συμβούλιο να μου εξηγήσει πώ θα είμαι βέβαια ότι μετά την αδειοδότηση εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας εάν δεν υπάρχει ε, αν δεν ε, διακυβεύεται τίποτα για την εταιρεία. Πώς θα την πείσω εγώ να με μεριμνήσει για την ασφάλεια. Αυτό λοιπόν πρέπει να μου το εξηγήσει το Συμβούλιο, αν έχει αντιρρήσεις. Θα γίνουν συστήσει λοιπόν με το Συμβούλιο, αλλά πρώτα πρέπει να συμφωνήσουμε στην Επιτροπή μα. Τι θέλουμε. Και πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε μαζί. Είναι ένα τεράστιο θέμα για τη δημόσια ασφάλεια και έτσι, ελπίζω αγαπητοί συνάδελφοι, αν μπορούσαμε από κοινού να συμφωνήσουμε στις τροπολογίες που μπορούμε να καταθέσουμε, να το πράξουμε από κοινού για να προχωρήσουμε ταχύτερα και έτσι να συνάψουμε τις συζητήσεις, να αναλάβουμε τις συζητήσεις με το Συμβούλιο ε, πολύ νωρί για να είμαστε έτοιμοι τον Ιούλιο για την ε, θέση σε ισχύ της νομοθεσίας. Και πρέπει να επισημάνω εγώ προσωπικώ ότι από αυτή όλη την ιστορία έχω διδαχθεί ότι χρειάζεται η σωστή φαρμακογρύπνευση στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί δεν μπορούμε να αρκούμαστε σε καλή νομοθεσία που θα ισχύει ενδεχομένω σε μία χώρα, γιατί μπορεί τα προϊόντα αυτά να κυκλοφορήσουν σε άλλε χώρε. Άρα χρειάζεται καλό και σωστό διάλογο και μεταξύ των κυβερνήσεων, μεταξύ των κρατών μελών και μια ενισχυμένη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μακέβαν. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ τους προσκεκλημένους μας που κάθονται πίσω προς τα παράθυρα. Είναι 37 ε, μαθήτρες του Γυμνασίου Ε, Τις έχει καλέσει εδώ τις μαθήτριες η συνάδελφος κυρία Μωρίν. Σας καλωσορίζουμε θερμά στην Επιτροπή μας και ελπίζω να απολαύσετε τις συζητήσεις που θα ακούσετε εδώ στην Επιτροπή μας. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα με τον κατάλογο των σκιωδών εισηγητών. Ε, Θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Πιλάρα Αγιούζο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, χαίρομαι πολύ που συνεργάζομαι και πάλι με την κυρία Μακάβαν και τους υπόλοιπους σκιώδεις που, προσπαθ... που είχαμε εργαστεί και για την τροποποίηση της προηγούμενες φορές ε, της οδηγίας και του κανονισμού για την ε, φαρμακοεπιτήρηση. Τα είπε τα περισσότερα νομίζω. Είναι μια ελάχιστη τροποποίηση μιας νομοθεσίας που μόλις τώρα αρχίζει να ισχύει. Σύμφωνα απόλυτα μαζί της να επιταχύνουμε πρέπει όλη τη διαδικασία ούτω ώστε όταν θα αρχίσει να ισχύει τον Ιούνιο του 2012 η νομοθεσία αυτή να έχει συμπεριλάβει τις ε, σωστές τροποποίησεις. Είναι αναγκαίες. Ακριβώς λόγω της υπόθεσης διατόρα. υπήρχε κενό, πρέπει να το καλύψουμε. Συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής. Σύντομα μπορούμε να καταλήξουμε, χωρίς προβλήματα. Δεν είναι σημαντικές οι αλλαγές. Η νομοθεσία πρέπει να αρχίσει να ισχύει εντελώς μεταρρυθμισμένη. Ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή τα δύο. Το πρώτο είναι το 123 του τμήματος 2 της οδηγίας όπου λέτε ότι αυτοί που έχουν την άδεια, οι αδειοδοτηθέντες, πρέπει να ενημερώσουν όλα τα κράτη-μέλη για οποιαδήποτε αλλαγή που γίνεται και που θα μπορούσε να προκαλέσει την αναστολή ή ανάγκη ανανέωση μιας άδειας. Θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή εάν είναι όντως αναγκαίο αυτό να ενημερώσει όλες τις χώρες ή μόνο τα κράτη-μέλη όπου έχει εγκριθεί το φάρμακο αυτό. Και όχι όπως προτείνει όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί ούτως ή άλλως το θέμα θα το δει η Επιτροπή Κινδύνων της Φαρμακοεπιτήρησης. Όλα τα κράτη-μέλη εκ των υστέρων θα το μάθουν. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ε, ε, υπερβολική διοικητική ευθύνη και φόρτος εργασίας για τα κράτη-μέλη και εφόσον πρόκειται για, για, κάποιο κράτος μέλος που δεν χρησιμοποιεί αυτό το φάρμακο, που δεν ε, κυκλοφορεί, για ποιο λόγο. Άλλη αμφιβολία. Για τις επίγουσε διαδικασίε που προβλέπονται στο 107, στο σημείο ε, λέει ότι αν υπάρχει μια νέα αντένδειξη, μια μείωση της δόσης, μια... ένας περιορισμός των λόγων για τον οποίο πρέπει να λαμβάνεται, πρέπει αυτόματα να προκαλεί επίγουσα διαδικασία. Και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων πρέπει σε ορισμένο χρονικό διάστημα να αρχίσει. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, αλλά θα ήθελα να μάθω γιατί χρειάζεται έτσι ακριβώς όπως διατυπώνεται αυτό το άρθρο. Συμφωνώ κατά τα υπόλοιπα εντελώς με αυτά που είπε η κυρία Μακάβαν. Ευχαριστώ. Πέτσα Λίζα. Και μετά Ανδρέα Ζανώνη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να στηρίξω όλα αυτά τα οποία είπαν οι δύο προλαλήσασες συνάδελφοι και νομίζω ότι δεν θα καταθέσω ε, τροπολογίες όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής. Ε, πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Θα ήθελα μόνο να εκφράσω δύο παρακλήσεις δικές μου προς την εισηγήτρια και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά λοιπόν την ποιότητα της ε, φαρμακοεπαγρύπνησης, η ποιότητα αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με το νομοθέτημα το οποίο συζητάμε. Εγώ θέλω να αναφέρω δύο θέματα τα οποία είναι σημαντικά, τα συζητάμε στο πλαίσιο άλλων οδηγιών και αφορούν στην ασφάλεια των φαρμάκων και στη βελτίωση αυτών και της φαρμακοεπαγρύπνησης. Στην αρχική λοιπόν πρόταση της Επιτροπής για την φαρμακοεπαγρύπνηση προβλεπόταν να υπάρχει είδος, ένα είδος κουτιού γεγονότων που θα συγκεντρώνονται δεδομένα για τα φάρμακα. Fact box, ας το πούμε έτσι. Αυτή λοιπόν η ε, πρόταση το Συμβούλιο απέτησε να διαγραφεί αλλά εμείς ε, μετά από συζητήσεις που είχαμε καταλήξαμε ε, στο ότι έπρεπε να αφήσουμε αυτή την πρόταση στην ε, έκθεση της κυρίας Μακάβεν και μετά στην έκθεση του κυρίου Κρίσοφα Κέλνουν για την ενημέρωση των ασθενών την επαναφέραμε την πρόταση αυτή. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει έτσι μια περίληψη των σημαντικότερων αντενδείξεων. Γιατί ξέρετε οι ασθενείς δεν διαβάζουν όλες τις οδηγίες που αναφέρονται στα φάρμακα. Ε, δεν θέλω βέβαια να επαναφέρω αυτή την τροπολογία, θα ήθελα όμως να παρακαλέσω όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους να μην προσποιούνται ότι εμείς ανέκαθεν ε, ήμασταν αντίθετοι. Όχι, κάθε άλλο. Και στη Φιέλνα και στην περίπτωση της πρώτης έκτης κύρια Μακάβαν συμφωνήσαμε. Όμως ε, το θέμα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω από την Επιτροπή και πρέπει με τον ενδεδειγμένο τρόπο να κάνουμε κι εμείς κάτι. Γιατί πράγματι βοηθάει το να έχουν έτσι κάποιο προσανατολισμό οι ε, ασθενείς και να μην είναι αναγκασμένοι να διαβάσουν όλες αυτές τις σελίδες που περιλαμβάνουν τα μικρά φυλάδια μέσα στις συσκευασίες ε, φαρμάκων. Κάτι άλλο τώρα. Η καταχώρηση των ε, κλινικών ερευνών. Ένα άλλο σημαντικό θέμα για την φαρμακοεπαγνήτηση ήταν για μένα το φάρμακο Vioxx ε, το οποίο ε, αποσύρθηκε λόγω σημαντικών επιπτώσεων στο ε, καρδιαγκιακό σύστημα. πολλοί είπαν ότι οι αντιδείξει ήταν ήδη γνωστέ πριν εγκριθεί το φάρμακο και κυκλοφορεί στην αγορά. Άρα δηλαδή δεν χρειάζεται να υπάρχει μεγαλύτερη φαρμακοπαγρύπνη στο μέλλον για να αποφευθούν παρεμφερεί περιπτώσει. Ότι αρκεί δηλαδή να καταχωρούνται όλε οι κλινικέ δοκιμέ. Γιατί αν είναι δυνατόν ορισμένα αποτελέσματα να μην δημοσιεύονται επειδή είναι αρνητικά, θα εμφανίζονται συνεχώ τέτοιου περιπτώσει και θα είναι και άχρηστη η φαρμακοεπαγρύπνηση. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ την Κομισιόν στην πρότασή τη για τι κλινικέ δοκιμέ να συμπεριλάβει και αυτή την πρόταση. Δηλαδή, όταν γίνονται κλινικές έρευνες σε τρίτες χώρες, να διασφαλίζουμε, να επαληθεύουμε ότι πράγματι αυτές λαμβάνουν χώρα και όχι αν τα αποτελέσματά τους είναι αρνητικά να αποκρύπτονται. Αυτά τα δύο θέματα ήθελα να θίξω. Θα ήθελα, ε, βέβαια, να μην επιβαρύνω την έκθεση της κυρίας Λίντα Μακέιβεν, θα ήθελα απλά να παρακαλέσω την Κομισιόν να μας πει κατά πόσο είναι πρόθυμη να τοποθετηθεί στις δύο άλλες ε, νομοθετικές διαδικασίες που τρέχουν παράλληλα. Ο κύριος ε, Τσανόνη και μετά η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, λαμβάνω και εγώ το λόγο εκ μέρου ε, των ε, φιλελευθέρων, εκ μέρου τη συναδέλφου κυρία Παράνοβα, Παράνοβα που δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα το πρωί. Η δική μα λοιπόν η ομάδα δέχεται και συμφωνεί τι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνεί επίση με την έκθεση τη εισηγήτρια. Μετά από αυτό το stress test το περίφημο του φαρμάκου Mediator, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει κενά που υπάρχουν στην νομοθεσία του 2011. Αυτά λοιπόν τα κενά πρέπει να αντιμετωπιστούν έτσι ώστε να μπορέσουμε να αγγιθούμε ένα βέλτιστο πλαίσιο για τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Επειδή λοιπόν εντοπίστηκαν όπως είπαμε κενά και στο μελλοντικό νομοθετικό πλαίσιο κενά τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την ασφάλεια των ασθενών είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε την, ε, όσο πιο, ε, την ταχύτατη έγκριση αυτής της ε, έκθεσης έτσι ώστε να ενταχθεί και αυτή στην νομοθεσία του 2011 και η δυνατόν να τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2012. Όσον αφορά τώρα την περίπτωση του φαρμάκου Mediator, έχουμε δικαστικές αποφάσεις κατά τι εταιρείε τη Σερβιέ. Αυτές οι αποφάσεις τρέχουν στη Γαλλία. Πρέπει όμως να περιμένουμε το αποτέλεσμα ε, των ερευνών. Καλύτερα λοιπόν να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτά που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να τηρούμε όλες τις αποφάσεις και προτάσεις τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τώρα το περιεχόμενο της πρότασης ε, της Επιτροπής, η ομάδα των φιλελευθέρων είναι ευνοϊκά διακείμενη απέναντι στα μέτρα που προτείνονται για να επικαιροποιηθεί ε, η βελτιστοποίηση της ε, νομοθεσίας, το άρθρο 107 συγκεκριμένα. Είναι λοιπόν νομίζω σκόπιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πράγματι απαραίτητο. Δηλαδή όταν μια εταιρεία αποφασίζει να αποσύρει ένα φάρμακο για λόγους ασφάλειας τότε η κατεπίγουσα διαδικασία πρέπει να ε, δρομολογείται, να ξεκινάει αυτόματα και αυτεπάγγελτα. Ε, πολύ ωραία. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ η υπόθεση αυτή με διατόρ που ξέσπασε στη Γαλλία είναι ενώπιον της δικαιοσύνης θα γίνει σίγουρα μια δίκη που θα έχει μεγάλη σημασία και κατόπιν μετά από αυτή την απόφαση τα τεστ αντοχής, stress test που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέδειξαν ότι υπήρχαν κενά Πρώτον, έλλειψη συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν ένα κράτο μέλο θέλει να αποσύρει, να αναστείλει ή να μην ανανεώσει μία αδειοδότηση κυκλοφορία και δεν θεωρεί ότι χρειάζεται επίγουσα δράση, δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση της ασφάλειας του προϊόντος σε επίπεδο ένωσης Πρέπει λοιπόν ο αυτοματισμός αυτής της ε, προειδοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι η μικρή μου διαφοροποίηση και μένα σε σχέση με τους συναδέλφους του ΕΛΚ. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει συνέπεια και ε, παρόμοια αντιμετώπιση ε, από όλα τα κράτη-μέλη, ακόμη και αν αυτό επιφέρει διοικητικές επιπλοκές, είναι σημαντικό όλη η Ένωση να δράσει. Το δεύτερο κενό, έλλειψη αιτιολόγησης από αυτούς που έχουν την άδεια και που το αφαιρούν, το, το αποσύρουν το προϊόν αυτό. Δεν είναι υποχρεωμένοι να εξηγήσουν γιατί το αποσύρουν. Με την αλλαγή που προτείνουμε θα πρέπει να αναφερθούν οι λόγοι. Απολύτως απαραίτητο πιστεύω. Για περισσότερη διαφάνεια. Τρίτο κενό. Έλλειψη αξιολόγησης μετά την αδειοδότηση. Έχουμε ένα κατάλογο προϊόντων, που, φαρμάκων δηλαδή που χρειάζονται συμπληρωματική επιτήρηση και ορισμένα φάρμακα χρειάζονται μια διαδικασία ελέγχου ασφάλειας και μετά την αδειοδότηση. Τι είναι λοιπόν σημαντικό, όπως είπε η κυρία Μακάβαν, είμαι πεπισμένη ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε όλοι για το θέμα αυτό πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Οι προθεσμίες είναι πολύ ε, προσεχείς, ούτως ώστε να υπάρξει διαφάνεια, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, αν υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια ενός φαρμάκου. Τώρα τον δημόσιο κατάλογο προϊόντων που είναι αντικείμενο ιδιαίτερης επιτήρησης μετά την αδειοδότηση, να επιλέξουμε σωστά τα φάρμακα αυτά που χρειάζονται ιδιαίτερη παρακολούθηση. Να μην δημιουργηθεί, καχυποψία στους ε, ασθενείς. Μετά την επίθεση Mediator είδαμε ότι οι διάφοροι ασθενείς δεν εμπιστεύονταν τα φάρμακα. Αυτό είναι καταστροφή για τη βελτίωση της υγείας και η πρόσβαση στην υγεία περνάει μέσα από την εμπιστοσύνη μεταξύ άλλων και προς τα φάρμακα. Καλύτερο λοιπόν πιστεύω να κάνουμε την αποτίμηση και αξιολόγηση ανά προϊόν και όχι να προτείνουμε έναν εκτεταμένο κατάλογο που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Πέρα από τα κενά που ε, επέδειξαν τα stress test της Κομισιόν, πρέπει να δούμε και τι, έγινε με τα, τι γίνεται με τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται χωρίς αδειοδότηση. για άλλες ενδείξεις θεραπευτικές και αυτή η χρήση προκαλεί ε, κλινικούς κινδύνους. Και σε αυτό το θεωρώ ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων να, αναλάβει, να αναπτύξει σε, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση εκτός ε, της ε, υποχρέωσης αυτής ώστε να διαφυλαχθεί η να εξασφαλιστεί μια ευελιξία για τις θεραπευτικές γραμμές ώστε να ικανοποιούνται και οι θεραπευτικές ανάγκες του κάθε ασθενούς. Αυτή η περίπτωση βέβαια του ε, Μεντιατόρ πρέπει να σας πω ότι εμένα με έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Με έχει προβληματίσει το θέμα της αδειοδότησης σε εθνικό, σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν υπήρχε μόνο ευρωπαϊκή αδειοδότηση, ίσως θα αντιμετωπίζαμε όλα τα θέματα πολύ πιο εύκολα. Ξέρω ότι δεν είναι η στιγμή να το θέσουμε αυτό, αλλά όταν εξασφαλίσει αυτή η εξέλιξη θα αντιμετωπίσουμε όλες, όλα τα προβλήματα. Σόλεμος και μετά Ήπνερ. Thank uh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες και τους λόγους για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει την πρόταση, γιατί βλέπω ότι είναι ξεκάθαρη στους πάντες οι λόγοι αυτοί. Έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα, έχουμε κάνει την ε, ανάλυση της κατάστασης και προσπαθούμε τώρα να κλείσουμε τα παραθυράκια. υπάρχουν ένα-δύο σημεία όπου θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρει περισσότερες εξηγήσει για, την, για τους λόγους που την οδηγούν στις προτάσεις της. Η ανάγκη για κοινοποίηση από την αδειοδοτηθεί σε εταιρεία, από τον αδειούχο δηλαδή, ε, περί μιας απόφασης ε, για διακοπή ή αναστολή απόσταση από την αγορά ενός προϊόντος. Πρέπει να κοινοποιήσει σε όλες τις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών. Και δεύτερον, γιατί αυτόματα η διαδικασία, η κοινοτική διαδικασία θα πρέπει να ε, τεθεί αυτόματα σε λειτουργία εάν υπάρχει περιορισμός ως προς τις ενδείξεις ή τις δόσεις. Πρώτο σημείο, κοινοποίηση προς όλα τα κράτη-μέλη. Μας απασχόλησε το θέμα αυτό, το μελετήσαμε προσεκτικά. Καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες είναι απαραίτητο όλα τα κράτη-μέλη ε, να βεβαιούμαστε ότι θα είναι ενημερώ όλα τα κράτη-μέλη. Και έστω και αν το συγκεκριμένο προϊόν δεν διατίθεται στην αγορά, μπορεί να υπάρχει ένα αντίστοιχο προϊόν, ένα παρόμοιο, με την ίδια δραστική ουσία. Για να μην δημιουργηθεί λοιπόν επιπλέον παραθυράκι, για να μην προσπαθήσει κανείς να αποφύγει έστω και την περιορισμένη αυτή ροή πληροφοριών, που ορισμένοι φαίνεται ότι θεωρούν όχι τόσο σημαντική από ό,τι ακούμε, ε, πιστεύουμε ότι το καλύτερο θα είναι να κλείσει κάθε κενό για να μην υπάρχει πρόβλημα, για να μην ξανααντιμετωπίσουμε δηλαδή τέτοια προβλήματα που θα προκύπτουν από κενά στην νομοθεσία σε μερικά χρόνια. Είναι απαραίτητο να γίνεται κοινοποίηση παντού. Και αν κάποιο κράτο μέρο θεωρεί ότι δεν το αφορά, το αντιμετωπίζει όπω θεωρεί. Πάντως το γεγονός ότι υπάρχουν προϊόντα ή δραστικές ουσίες που μπορεί να ανήκουν στην ίδια οικογένεια προϊόντων Φερρυπίν ή ότι μπορεί να υπάρχουν προϊόντα με αντίστοιχο τρόπο δράσης που έχουν ήδη ε, διατεθεί στην αγορά, θεωρούμε ότι είναι σωστό, είναι απαραίτητο και ότι δεν έχει άμεση συνάφεια με το συγκεκριμένο φάρμακο ή προϊόν να γίνεται κοινοποίηση σε όλες τις αγορές, σε όλες τις χώρες. Γιατί είναι αυτόματη διαδικασία, όταν εμφανίζονται νέε αντεδείξει ή περιορισμοί προ τι ενδείξει. Οι δράσει που προβλέπονται, εφόσον είναι για λόγου ασφάλεια, μπορεί να ε, οφείλονται σε πολύ σημαντικές ε, επενέργειες και ως εκ τούτου για να μην έχουμε σε λίγο πάλι πρόβλημα λόγω κάποια ουκενού στην νομοθεσία, λέμε ότι δράσεις που έχουν να κάνουν με την ανησυχία για λόγους ασφάλειας πρέπει να ισχύουν σε όλη την Ευρώπη για να είμαστε σίγουροι ότι οι πάντες στηρούν τους ίδιους κανόνες. Αυτή είναι που αυτά τα σημεία που βλέπουμε ότι χρειάστηκε να δώσουμε κάποιες εξηγήσει. Πέραν αυτού σημειώνω την υποστήριξη που εκφράζει η Επιτροπή σας στις ε, προτάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν να δώσω το λόγο για να καταλήξει την, ε, καταλήξει την συζήτηση, να ενημερώσω τους Δανούς συναδέλφους ότι έχουμε και πάλι Δανέζικη καμπίνα. Δίνω το λόγο στην Λίντα Μακάβαν να μας πεις Λίντα παρακαλώ πότε θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή 8 ή 30 Μαΐου γρήγορα ή όχι τόσο γρήγορα για την ε, ημερομηνία ακούγοντας τους συναδέλφους νομίζω ότι επειδή έχουμε μια άλλη συνεδρία των συντονιστών την άλλη εβδομάδα αν χρειάζεται οποιαδήποτε αλλαγή μπορούμε λοιπόν τότε αλλαγή στην πρόταση της Επιτροπής μπορούμε να το αποφασίσουμε τότε θέλω να είμαι σίγουρη ότι η εταιρεία πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι δεν απέσυρε το φάρμακο για λόγους ασφαλείας. Γιατί στην περίπτωση ενδιατόρι είπαν ότι ήταν για εμπορικούς λόγους. Ξέρετε, αυτή είναι νομική συζήτηση. Θέλω να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μπορούν να λένε κάτι που όλοι θα ξέρουμε ότι δεν ισχύει. Θέλω να ελέγξω τη διατύπωση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ουσίας δεν νομίζω ότι έχουμε να προτείνουμε αλλαγέ στην πρόταση της Κομισιόν. Να υποβάλω την πρότασή μου πριν το Πάσχα για να μεταφραστεί και ίσως θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε στις 8 Μαΐου. Όσο συντομότερα ψηφίσουμε, τόσο συντομότερα μπορούμε να αρχίσουμε το διάλογο με το Συμβούλιο. Ξέρω ότι έχει κάποιες ανησυχίες, μπορεί να μην πάει τόσο γρήγορα η διαδικασία. Γιατί θέτουν κάποια ερωτήματα για το μαύρο τρίγωνο, την ε, έντονη επιτήρηση. για το θέμα γιατί όλα τα κράτη-μέλη και όχι μόνο εκεί που κυκλοφορεί, που ανέφερε η κυρία Γιούσο. Αλλά αν μια χώρα το αποσύρει εθελουσίω σε μια χώρα, αν μια εταιρεία το αποσύρει εθελουσίω σε μια χώρα και όχι σε άλλε. δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Ναι, ναι, μπορεί διοικητικά να είναι κάπως πιο βαρύ, αλλά όλοι θα έχουν την πληροφόρηση και κανεί δεν θα μπορεί να πει ότι δεν ήξερα. Ξέρω ότι στη συζήτηση γίνεται πολύ συζήτηση για το θέμα. στο Συμβούλιο γίνεται πολλή συζήτηση για το θέμα αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο σοβαρό για την επίγουσα διαδικασία. Η διατύπωση της Επιτροπής μιλάει για λόγους ασφαλείας. Ξέρουμε ότι ορισμένα φάρμακα μπορεί να αποσυρθούν για εμπορικούς λόγους, γιατί δεν πουλάνε. Δεν θέλουμε όλη αυτή την επίγουσα διαδικασία, αν ειλικρινά όντω είναι για εμπορικού λόγου. Να πούμε ότι η επίγουσα διαδικασία σχετίζεται με θέματα ασφάλεια. Σκόπιμο. Γιατί αν το αφήσουμε στη διακριτική ευχέρεια των εταιριών, όπω το Mediator, έγιναν άτυπες συζητήσεις, αλλά δεν υπήρχε υποχρέωση συζήτησης να μην ξανασυμβεί. Για αυτά που είπε το περίφημο μαύρο κουτί. Δεν ξέρω τι έγινε σε αυτή την επιτροπή. Το συζητήσαμε και το είχε υποστηρίξει εγώ το μαύρο κουτί. Στρέφομαι και προς τους άλλους ε, σκιώδεις. Είχαμε πολύ, πολλές οργανώσεις ε, ασθενών που μας έλεγαν ότι δεν συμφωνούν όλοι για το τι είναι σημαντικό και τι όχι. Ρωτήσαμε και την Επιτροπή. Ίσως όχι ενδεχομένως σήμερα, να μας πει η Επιτροπή, γιατί νομίζω ότι το φυλάδιο η ενημέρωση των ασθενών θα ε, το επανεξετάσουν και ίσως θα το επανυποβάλουν φέτος ή του χρόνου. Όταν λοιπόν το επανεξετάσετε, όταν θα μας κάνετε πρόταση γι' αυτό, σας υπενθυμίζουμε να μας υπενθυμίσετε πότε θα υποβάλλετε αυτή την νέα εκδοχή του. Για τις ε, κλινικές δοκιμές υπάρχουν άλλοι πιο εμπειρογνώμενες από μένα για αυτά που είπε η κυρία Γκροστέτ για το μαύρο τρίγωνο. Έχει δίκιο. Δεν πρέπει να φοβίζουμε τους ασθενείς για τα φάρμακα. Αλλά αυτή τη στιγμή μειώνεται η εμπιστοσύνη του κοινού. Είχαμε αυτή την περίπτωση. Είχαμε την περίπτωση με τα εμφυτεύματα. Ναι βεβαίω και αυτή η γαλλική υπόθεση. Αλλά έχουμε τώρα ένα θέμα με τα εμφυτεύματα ισχύων το κοινό δεν είναι και τόσο ε, ικανοποιημένο από τις κανονιστικές μας διαδικασίες. Αν θέλουμε λοιπόν να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη, κάτι πρέπει να κάνουμε. Υποστηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο. Είπατε ότι οποιοδήποτε φάρμακο που χρειάζεται μελέτη μετά την αδειοδότηση για την ασφάλεια πρέπει να φέρει αυτό το μαύρο τρίγωνο μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη. Αυτό το υποστηρίξαμε κι εμείς το Συμβούλιο μας πίεσε πολύ και το αποδεχθήκαμε και η Επιτροπή το αποδέχθηκε. Αλλά εγώ το ξανασκέφτηκα. Δεν κάναμε καλά που υποχωρήσαμε. Θα πρέπει να μείνουμε στην αρχική μας πρόταση. Μπορούμε να δούμε σε πόσα φάρμακα θα το εφαρμόζαμε. Αλλά θέλουμε οι ασθενείς να είναι ενημερωμένοι και υπόθηκε ότι το να πάρει κανεί ένα φάρμακο είναι όφελος, είναι και ρίσκο. Γιατί υπάρχουν πάντα παρενέργειες. Το μαύρο τρίγωνο υποχρεώνει τον ασθενή να εξηγήσει στον, υποχρεώνει τον ιατρό να εξηγήσει στον ασθενή τι συμβαίνει και όχι απλώς να το γράψει. Θέλουμε λοιπόν ενημερωμένους ασθενείς ούτω ώστε να συμμετέχουν μαζί με του επαγγελματίε τη υγεία στην φάρμακο επαγρύπνηση. Δεν θέλουμε μια φαρμακευτική εταιρεία μια μελέτη που έπρεπε να την κάνει ένα χρόνο να την κάνει 8. Δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Εγώ νόμιζα ότι πάντα γίνονται μελέτε και ότι όλοι δρούν υπεύθυνα, αλλά πρέπει να το διασφαλίσουμε αυτό. Ακούσαμε το θέμα για τη χρήση χωρίς ετικέτες νομίζω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται αυτό. Δεν θα ήθελα να σταματήσει Δεν θα ήθελα να σταματήσει η, η χρήση χωρίς εργαστήρια. Χωρίς να έχουμε δοκιμές από τα εργαστήρια. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει παρακολούθηση από την κυβέρνηση και από τους επαγγελματίες της υγείας και η κυβέρνηση ελέγχει τον τρόπο συνταγοδότησης. Για παράδειγμα για θέματα δυνατίσματος. Σε αντιδιάσταση με, την, με τον διαβήτη έπρεπε να το έχουμε εξετάσει. Αλλά δεν ξέρω αν έχει έννοια τώρα να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση για την συνταγοδότηση χωρίς κλινικές δοκιμές, χωρίς εργαστηριακές δοκιμές. Είπαμε επίσης ότι η ανείχνευση των ε, ε, ε, η ανείχνευση των απόψεων και των πληροφοριών που έχουν οι, ασθεν... ιατροί όταν ένα ασθενή του πει ότι πήρα αυτό το φάρμακο και είχα αυτέ τι παρενέργειε. Θα πρέπει λοιπόν όλη αυτή η πληροφόρηση να μπαίνει σε τράπεζε δεδομένων. Μια άλλη αλλαγή που κάναμε είναι ότι βελτιώσαμε πολύ την ενημέρωση του κοινού για τις αντενδείξει. Πρέπει φυσικά οι ασθενεί να παίρνουν φάρμακα, αλλά να τα παίρνουν ενημερωμένα. Και ότι κλείσαμε όλα τα παραθυράκια που μπορεί να υπονομεύουν την ασφάλεια των φαρμάκων. Πρόεδρος. Πίτσα Λίζε. Σύντομη συμπληρωματική ερώτηση στην Επιτροπή και μία διευκρίνηση. Γι' αυτό το κουτί για, μεταδεδομένα Στην πρόταση της Επιτροπής για τη φαρμακοεπαγρύπνηση πριν από 2-3 χρόνια, το 2008, αυτό το μαύρο κουτί, το κουτί με τα στοιχεία προβλεπόταν, έγινε μια συζήτηση και εγώ είπα δεν πρέπει να είναι μαύρο κουτί, δεν χρειάζεται να είναι αυτού του τύπου το μαύρο κουτί, μπορούσε να γίνει και αλλιώ. Αλλά η Επιτροπή μας δεν ενέκρινε την διαγραφή του. Σωστά είπε η Λίντα, υπήρξαν επικρίσεις, αλλά εγκρίναμε χωρίς τροποποίησης την πρόταση της Κομισιόν. Μετά στον τρίλογο, λόγω ποιήσης του Συμβουλίου το διαγράψαμε. Αλλά όπως είπαμε ήταν η συμφωνία για την πρώτη ανάγνωση. Αλλά κανείς δεν ήθελε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ήμασταν κατά. Στην Επιτροπή δεν εγκρίναμε τροπολογίες, εγκρίναμε ατροπολόγητη την άποψη της Επιτροπής και κατόπιν από τον, από τον τρίλογο διαγράφει. Και τότε μετά εγκρίναμε την έκθεση Φιέλνερ για την μέρος των ασθενών, όπου η πλειοψηφία στην Ολομέλεια, στην πρώτη ανάγνωση, αποφάσισε ότι το θέλουμε αυτό το κουτί. Μπορούμε όλα να τα ξασυζητήσουμε, αλλά να μην μπούμε ότι ήμασταν κατά του κουτιού αυτό. Να μου πει λοιπόν η Επιτροπή, αν αυτή την πρόταση της έκθεσης Φιέλνερ ή κάπου αλλού θα την συμπεριλάβει. Ή αν πρέπει να κάνουμε μια τροπολογία για να συζητηθεί και πάλι το θέμα αυτό, αλλά δεν θα το ήθελα. Η διαδικασία για την έκθεση τη Λίντα δεν πρέπει να επιβαρυνθεί και με το θέμα αυτό. Κανεί να μην πει όμω ότι το Κοινοβούλιο είναι κατά του κουτιού. Εμεί είμαστε υπέρ του κουτιού. Και κάτι άλλο τώρα. Θεωρεί η Επιτροπή ότι πρέπει να εξετάσει να υπάρξει ένα μητρό των κλινικών δοκιμών στα πλαίσια της ε, σχετικής οδηγίας. Αυτό θα μας βοηθούσε να βελτιώσουμε τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Ίσως δεν ε, πρέπει να το βάλουμε στην πρόταση τώρα, μακάβαν, αλλά θα μπορούσαμε σύντομα να το συμπεριλάβουμε. Εάν έχουμε την πολιτική κατεύθυνση της Επιτροπής για αυτό. Ευχαριστώ. Λίζε. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Η Φρασουάζ Προχωριστέτ, μια συμπληρωματική ερώτηση. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είχα θέσει ένα ζήτημα το οποίο μου φαίνεται πολύ σημαντικό. Καταρχάς, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στην Γαλλία ο Υπουργό Υγεία αποφάσισε ήδη ε, κάποιε τροποποίησεις στην εθνική νομοθεσία για τη φαρμακοεπαγρύπνηση και έτσι ε, ορίζει πιο αυστηρούς ε, κανόνες, πιο αυστηρές διατάξεις. Ε, ύστερα από αυτή την γενική συζήτηση για τα φάρμακα, τη συνέλευση των φαρμάκων, τη οποία είμαι και εγώ μέλο, Αλλά θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή για άλλη μια φορά σε σχέση με την χρήση του φαρμάκου εκτός AMM. Και θέλω να ρωτήσω εάν μπορούμε να στήσουμε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων σε συνεργασία με τις Εθνικές Υπηρεσίες να εκπονήσει για το off-label use των φαρμάκων, την χρήση δηλαδή Εάν μπορεί να αποφασίσει λοιπόν να ρυθμίσει το ζήτημα κατά αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει για άλλη μια φορά το λόγο για να δώσει απαντήσει στι ερωτήσει που έχουν του μεταξύ τεθεί και τι ε, συστάσει των, προτάσει των συναδέλφων. Παρακαλώ. Πρόεδρε. Το μαύρο κουτί. Θα ήθελα καταρχά να επισημάνω, να διευκρινίσω ότι η πρόταση που έχουμε έχει σαν στόχο να προσδιορίσει, να εντοπίσει και να ρυθμίσει αδυναμίες του συστήματος που εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση, κατά το stress test δηλαδή. Και είπαμε ότι ήταν επίγον να αντιμετωπιστούν αυτά, εξού και κατατέθηκε πολύ γρήγορα μετά τον εντοπισμό των προβλημάτων η σχετική πρόταση. Εντοπίζουμε λοιπόν τα προβλήματα και τα ρυθμίζουμε, επιδιώκουμε τουλάχιστον να τα αντιμετωπίσουμε σε σχέση με την ε, προηγούμενη διαδικασία της συναπόφασης. Και τόσο έλαβαν χώρα εκεί. Έχω να πω ότι σε σχέση με το δελτίο ενημέρωσης του ασθενούς είναι η υποχρεωτική έκδοση μια έκθεση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναγνωσιμότητα του σχετικού αυτού φύλου, του φύλου ενημέρωση. Αρχίσαμε να αναλύουμε το πρόβλημα και όταν ολοκληρωθεί αυτή η ανάλυση θα είμαστε σε θέση εκ μέρους της Επιτροπής να καταθέσουμε έκθεση. Τι είδου πορίσματα θα βγουν από την έκθεση αυτή δεν μπορώ βέβαια να το ε, προεξοφλήσω τώρα, αλλά σας διαβεβαιώ και σας καθησεχάζω εφόσον χρειάζεται ότι ε, επεξεργαζόμαστε το θέμα. Όσον αφορά δε τις κλινικές δοκιμές, συζητούμε, επεξεργαζόμαστε ε, νέα πρόταση για κλινικές δοκιμές. Τώρα είμαστε στην ανάλυση επιπτώσεων. Έχουμε ένα δημόσιο μητρό όπου όλες οι κλινικές δοκιμές ε, υποχρεωτικά καταγράφονται και σε ένα βαθμό καλύπτονται πιστεύω όποιες ανησυχίες έχουν επισημανθεί. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Το ε, off-label ε, use σε ένα βαθμό ξεφεύγει από το πλαίσιο αυτής της πρότασης, δηλαδή μπαίνει ουσιαστικά στο χώρο της ιατρικής πρακτικής και θα δούμε πώς θα το χειριστούμε. για να ετοιμάσουμε δε η πρόταση για κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων. Προς το παρόν δεν μπορώ να δώσω απάντηση, γιατί είναι κάπως πρόωρο αυτό το έτοιμο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η έκθεση Μακέβαν, λοιπόν, θα συζητηθεί στην Επιτροπή μας 25 και 26 Απριλίου. Θα έχουμε τιμή και την μετάφραση με προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών την 27η Απριλίου. Και αν κατάλαβα καλά την κυρία Μακέβαν και τους λοιπούς ε, συναδέλφους και οδησηγητές, στις 8 Μαΐου θα πρέπει να ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας για να είμαστε έτοιμοι για την Ολομέλεια τον Ιούλιο. Ευχαριστώ θερμά την Επιτροπή για τις απαντήσεις της και τη συμμετοχή της και τώρα περνάμε στο σημείο 20 της ημερήσιας διάταξης όπου έχουμε συζήτηση με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, Διακρατική Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, σχετικά με την Παγκόσμια Οικονομική Συσμαστική Πράξη, σχετικά με τον Ιδράργυρο. Παρακαλώ, εκ μέρους της Επιτροπής. Καλημέρα σας. Και ευχαριστώ, Πρόεδρε, που δείτε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς ε, την ε, Επιτροπή σας για την ευκαιρία που μας δίνει να έρθουμε σήμερα και να σας εξηγήσουμε σε ποιο βαθμό έχουν προχωρήσει αυτές οι διαπραγματεύσεις για την ε, σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας δεσμευτικής για τον Ιδράργυρο από το το πρόγραμμα για το περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών και το σχετικό Διοικητικό Συμβούλιο. Μια απόφαση που είχε λεφθεί το 2009 αποτελεί το, την αφετηρία αυτή τη υπόθεση. και αποφασιστεί δηλαδή από την UNAP ότι είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα το θέμα του υδραργύρου και ύστερα από ε, προβλήματα για πολλά χρόνια κατέστη δυνατή σύναψη μια συμφωνία ω προ την ανάγκη για τη θέσπιση ενό νομοθετήματο παγκοσμίου ε, εμβέλεια για τον ε, υδράργυρο. Και δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 218 ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει να εκπροσωπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύσει. Είναι η πρώτη φορά όπου μπορούμε να προβούμε σε μια ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σα που μα καλέσατε. Σα ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μα δίνετε και θα ήθελα να εξηγήσω σε ποιο σημείο έχουν φτάσει οι συζητήσει αυτέ, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τι μένει ακόμη να γίνει στο μέλλον. Με στόχο την έγκριση του σχετικού νομοθετήματος. Στην απόφαση του 2002 του Διοικητικού Συμβουλίου είχε αποφασιστεί ότι θα γίνουν πέντε γύροι διαπραγματεύσεων από το 2010 έως το 2013 για τη συζήτηση του θέματος του υδραργύρου και ότι στη συνέχεια η διεθνή κοινότητα θα ήταν σε θέση πλέον να συνάψει αυτήν την διεθνή συμφωνία. Τρεις γύροι διαπραγματευτικοί έχουν λάβει χώρα μέχρι τώρα από τον Ιούνιο του 2010, ο πρώτος στη Στοκχόλμη, με τελευταίο τον ε, γύρο του Φεβρουαρίου 2013. που θα ακολουθήσει η ε, συνήθις διπλωματική διάσκεψη για την υπογραφή που προβλέπεται για το 2013 στην Ιαπωνία. Και γιατί στην Ιαπωνία, διότι η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, η οποία ήδη έχει φιλοξενήσει έναν ε, γύρο διαπραγματεύσεων, θέλει η διάσκεψη αυτή να λάβει το όνομα διάσκεψη Μιναμάτα από το όνομα της Ιαπωνικής πόλης Μιναμάτα, στην οποία έχει εμφανιστεί η χειρότερη περίπτωση ρήπανσης από υδράργυρο στην ιστορία της ανθρωπότητας πριν από 50 χρόνια και. Μετά τον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων στο Στοκχόλμη, ο δεύτερος ήταν το Φεβρουάριο του 2011 στην Ιαπωνία, στην Τζίμπα, ο τρίτος στο Ναϊρόμπι, τον Νοέμβριο του 2011 και τώρα ετοιμαζόμαστε για τον τέταρτο, τον Ιούνιο εφέτος, από 27 Ιουνίου μέχρι 2 Ιουλίου στην Πούντα Τελέστα της Ουρουάης. Έξι μέρες θα κρατήσει αυτή η συνεδρίαση, δηλαδή μια μέρα περισσότερο από ό,τι προηγούμενες, με στόχο τα θέματα ουσίας που έχουν εγγραφεί σε αυτέ τι διαπραγματεύσει να συστηθούν σε μικρότερου κύκλου συζητήσεων, όχι στην Ολομέλεια δηλαδή με παρούσε όλες όλε τι χώρε, πριν να υποβληθούν για συζήτηση στην Ολομέλεια. Και στόχος αυτού του τέταρτου γύρου ε, διαπραγματεύσεων είναι να εξασφαλιστεί συμφωνία για τα περισσότερα εκ των τμήματων που έχουν ήδη εντοπιστεί για αυτή την μελλοντική διεθνή συνθήκη. Πρέπει όμω να επισημάνω ότι μέχρι στιγμής λίγα μόνο ζητήματα έχουν επιληθεί. Ε, το πρόγραμμα λοιπόν, ε, ο σχεδιασμός όμως λέει ότι για τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα ο στόχος είναι να περιοριστούν οι, διαπραγμα... οι πληστηριασμοί μέχρι στον αριθμό που είχαμε μέχρι τώρα και να εξασφαλίσουμε μια συμφωνία. Και έχουμε εμείς ως βάση διαπραγματευτική την απόφαση των, μέσα από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου 2008 με στόχο την εξέταση ολόκληρου του βιολογικού κύκλου του υδραργύρου και τη λήψη των αποφάσεων με βάση αυτών. Έχουμε λοιπόν διάφορες ομάδες θεματολογικές που θα πρέπει να συζητηθούν στις ομάδες επαφής όπως το ονομάζουμε. Έχουμε την προμήθεια και το εμπόριο σε υδροόρκυρο και προϊόντα αυτού, τα προϊόντα και τις διαδικασίες παραγωγής, τη βιοτεχνία ή την, τα, τα μικρά χρυσορυχεία εκκλήσεις, εκπομπές υδραργύρου, αποθήκευση, απόβλητα και μολυσμένες τοποθεσίες και οικονομική πόρη, χρηματοπιστωτική πόρη και τεχνική στήριξη, δηλαδή αυτά είναι τα κεφάλαια στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Σε ορισμένα από αυτά τα θέματα, στους προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων έχουν συμμετεί σημαντικές πρόοδοι, ε, παραδείγματι στο θέμα των αποβλήτων ή επί στη χρήση του υδραργύρου στην ε, χρυσορυχία. Πλην όμως άλλα θέματα ακόμη δεν έχουν καν ε, αρχίσει να συζητούνται όπως είναι η προμήθεια ή το εμπόριο σε υδράργυρο. Ένα κύριο ζήτημα που ακόμα μένει να συζητηθεί, αναμφίβολα, είναι η χρηματοπιστωτική, η χρηματοοικονομική βοήθεια. Προφανώς αδίποτε λύση επιλαγή και μεταφραστεί σε μια μελλοντική συνθήκη για θέματα χρηματοοικονομικής ενίσχυσης θα πρέπει να είναι και συνεπής ως προς την προσέγγιση για τη χρηματοοικονομική ενίσχυση που έχει ληφθεί σε άλλες πολυμερείς περιβαλλοντικού χαρακτήρα συμφωνίες. Δεν μπορεί να έρχεται σε αντίφαση με αυτές. Ένα άλλο επίσης σημαντικό θέμα, πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πρόκειται για τεράστια πηγή παγκόσμιων, της παγκόσμιας ρήπανσης, είναι οι εκπομπές υδραργύρου στην ατμοσφαίρα, στον ατμοσφαιρικό αέρα. Έχουμε λοιπόν μια πολυμερή προσέγγιση με χρήση των βέλτιστων υφισταμένων τεχνολογιών. Η δε ευρωπαϊκή πλευρά θα πιέσει ώστε η προσέγγιση των βέλτιστων τεχνολογικών δυνατοτήτων να καταστεί υποχρεωτική μέσα στο τελικό κείμενο της συνθήκης. Η προσέγγιση αυτή δηλαδή ξέρουμε ότι μπορεί να αμφισβητηθεί από ορισμούς, εταίρους ε, στις ε, πραγματεύσεις αυτές, αλλά θα προσπαθήσουμε να τους πείσουμε ότι η βέλτιστη τεχνολογική προσέγγιση ή η τεχνολογία ως προσέγγιση μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα, είναι πρακτικά εφαρμόσιμη και άρα μπορεί να ε, εγκριθεί. Άλλα ζητήματα μένουν ακόμα να συζητηθούν, έχουν μείνει κάποιες λεπτομέρειες, πρέπει να συζητήσουμε. Στον τέταρτο επερχόμενο τέταρτο γύρο των διαπραγματεύσεων, θα πούμε στην πιο ουσιαστική φάση αυτών. Και κατά την προετοιμασία αυτού του γύρου των διαπραγματεύσεων πρέπει να σας πω ε, προχωρούμε αυτή τη στιγμή σε διατομιακή, ε, διατομιακή όπως τα λέγαμε, ή μάλλον ενδιάμεση δουλειά, δηλαδή στις περιόδους μεταξύ των διαφόρων συνόδων. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Έχουμε ε, συναντήσει στη Βουδαπέστη μεταξύ και 12 Απριλίου για το θέμα αυτό από ευρωπαϊκής πλευράς και αναλόγως του τι θα προκύψει εκεί θα δημοσιευθεί το νέο σχέδιο κειμένου για το νομοθέτημα για τον υδράργυρο στην ε, ιστοσελίδα της UNEP, του Προγράμματος των Εθνών για το Περιβάλλον. Και αυτό θα αποτελέσει τη βάση, σε προ, αυτού του Φεβρουαρίου, ε, θα αποτελέσει τη βάση ε, εργασίας. Έτσι λοιπόν αυτή η ενδιάμεση δουλειά που γίνεται στην Βουδαπέστη συμπληρώνεται και από άλλες δραστηριότητες για την προετοιμασία του επίσημου γύρου διαπραγματεύσεων που θα λάβει χώρα τον Ιούνιο οι διαπραγματεύσει λοιπόν αυτέ, οι μάλλον δραστηριότητε αυτέ, έχουν να κάνουν με μια συζήτηση για τι διαδικασίε που θα υποδεχθεί στο Τόκιο στο τέλη του Απριλίου η Ιαπωνία, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με άλλε σημαντικέ ε, ομάδε ή ε, χώρε, ομάδε χωρών ή χώρε, θα προσπαθήσει να εντατικοποιήσει ανταλλαγέ με άλλου εταίρους για να εξασφαλιστεί μια κοινή αντίληψη του ποιε είναι οι προκλήσεις που παρουσιάζει ο υδράργυρος και τα προϊόντα αυτού. Ως προς την εσωτερική προετοιμασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τέταρτο αυτό γύρο διαπραγματεύσεων, και συζητήσεων. Έχουμε συζητήσεις στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου, ομάδα εργασίας για διεθνή περιβαλλοντικά θέματα δηλαδή, και θα ε, γίνουν δύο συνεδριάσεις ειδικά για τον Ιδράργυρο ε, μέχρι τα μέσα Ιουνίου οι οποίες ακολουθούν προηγούμενες συνεδριάσεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Επιπλέον αυτών των τακτικών συνεδριάσεων ε, της ομάδας εργασίας θα, γίνει και μια πιο, θα γίνουν και κάποιες πιο ειδικέ ε, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα, 20 6 με 28 ε, Μαρτίου και άλλη μία στην Κοπενχάγη, η, μία, ε, εδώ, η πρώτη στις Βρυξέλλες, η άλλη στην Κοπενχάγη και πιστεύουμε ότι αυτές οι ειδικέ συνεδριάσεις θα διευκολύνουν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα την εξοπλίσουν για την ε, Ουρουγουάη με καλύτερα διαπραγματευτικά όπλα από ό,τι στο παρελθόν. Επιπλέον αυτό. Σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τις ανταλλαγές και την επικοινωνία με τους λοιπούς εταίρους, ώστε να είναι γνωστές οι θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και πριν από τις διαπραγματεύσεις ακόμη και να προσπαθήσουμε βέβαια και από πλευρά μα να αντιληφθούμε καλύτερα τι θέσει των λοιπόν σημαντικών διαπραγματευτικών μα εταίρων. Αυτή είναι η κατάσταση προ το παρόν. Βεβαίω και θα σα θυρούμε ενήμερου και θα, έρθουμε και θα σας αποστείλουμε γραπτός ενημέρωση μετά τον προσεχή γύρω διαπραγματεύσεων. Είμαι και εγώ και οι συναδελφοί μου στη θέση σας για οποιαδήποτε παρατήρηση ή ερώτηση που θα είχατε ενδεχομένω αυτό το στάδιο. Σα ευχαριστώ θερμά που μας δίνετε την ευκαιρία, που δώσατε την ευκαιρία να σας εξηγήσουμε την εξέλιξη διαπραγματεύσεων αυτέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Άννα Ρόσμπαχ. Ευχαριστώ με εκλέγουν πολίτες. Έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν για αυτή την πολύ επικίνδυνη ουσία. Δυστυχώς, ο υδράργυρος ε, είναι συστατικό πολλών προϊόντων που χρησιμοποιούμε στην, ε, χρησιμοποιούμε στην ε, καθημερινή μας ζωή που δεν τα περιμέναμε. Για παράδειγμα, οι κονσέρβες τόνου και σολομού. Οπότε, Πώς μπορούμε στην πράξη να μειώσουμε την έκθεσή μας στον υδράργυρο για τη φύση, τα άγρια ζώα και τους ανθρώπους. Όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Κίνα και την Ινδία που δεν συμμετέχουν σε αυτή την διαπραγμάτευση. Και πόσο θα κόστιζε στην, ε, πόσο κοστίζει στην οικονομία μας η διαρροή ε, υδραργύρου στη φύση αλλά και η επαφή που έχει στους ανθρώπους. Και θα ήθελα να μάθω εάν ε, εξορίγνεται στην Ευρώπη συνολικά ο υδράργυρος και πώς προστατεύουμε τους εργαζόμενους εάν ναι. Τελευταία ερώτηση. Δεν υπάρχουν άλλες ουσίες για να αντικαταστήσουν τον υδράργυρο. Και πάλι όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά γενικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκροστέτ. Και μετά ο κύριος Ζήμπα. Ευχαριστώ. Υπάρχουν διάφορες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία που είναι κατά των δεσμευτικών ε, αποφάσεων για την ε, μόλυνση από υδράργυρο. Νομίζω λοιπόν ότι είναι δύσκολη η δυνατότητα δράσης για τους οικονομικούς μηχανισμούς. Πολύ απέχουμε από μια συμφωνία για το θέμα αυτό τίθενται διάφορα ερωτήματα. Γιατί υπάρχει ανάγκη να συνεχίσουμε την ε, χρήση σε εξαιρετικές καταστάσεις του υδραργύρου για κάποια προϊόντα και διαδικασίες. Πώς μπορούμε να ορίσουμε λοιπόν τα όρια της χρήσης αυτής της κατεξαίρεση. Όσον αφορά τώρα την ε, αντιμετώπιση του υδραργύρου, δεν μπορεί να καταστραφεί. Πρέπει κάπου να αποθηκευθεί. Αυτό δημιουργεί προβλήματα. Είναι περίπλοκη η αποθήκευση και μεγάλο το κόστος. Αναμφίβολο. Και πώς αντιμετωπίζουμε την ε, εξαγωγή υδραργύρου. Θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιες μικρές ε, απομονωμένες περιοχές για την ε, αποθήκευση. Πώς θα χρηματοδοτήσουμε αυτή την προσπάθεια και τελευταίο, υπάρχουν κράτη που συνεργαζόμενα μεταξύ τους έχουν υιοθετήσει δεσμευτικά μέτρα. Για παράδειγμα, η Γαλλία και η, και η Βραζιλία μαζί καταπολεμούν την έκκληση υδραργύρου στην περιοχή του Αμαζονίου Συνεργάζεται λοιπόν εκεί η Γουιάννα, η Γαλλία και η Βραζιλία. Θα μπορούσε να υπάρξει και συνεργασία άλλου τύπου επίσης ε, θεσμευτική όπως αυτή που υπάρχει μεταξύ ε, Βραζιλίας και Γαλλίας. Ευχαριστώ πολύ Ζέμπετ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε η Επιτροπή. Αλλά λίγο είναι το περιεχόμενο όσον αφορά και τα, τα μέτρα και το, τις ποσότητες. Είναι πολύ επικίνδυνη λοιπόν αυτή η ουσία. Θα ήθελα λοιπόν να μας δώσει στοιχεία η Κομισιόν. Πώς θα μπορούσαν να επενεργήσουν αυτές τις στρατηγικές. Να μας πει η Κομισιόν πόσος υδράργυρος υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, πόσος παγκοσμίω, πόσος ετησίω και μία εκτίμηση για το πώς μπορούμε μακροπρόθεσμα να δράσουμε ούτως ώστε να καταργήσουμε εντελώς από την παραγωγή αυτό το προϊόν, ιδιαίτερα από την παραγωγή ενέργειας. Συγκεκριμένη ερώτηση. Πώς θα υποστηρίξουμε την έρευνα ούτω όταν να υπάρξουν οι αναγκαίε καταστάσει φιλτραρίσματο για να μην εκλείεται στο περιβάλλον. Τι εναλλακτικέ λύσει υπάρχουν στη χρήση του υδραργύρου. Στα ορυχεία είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η χρήση και το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος ε, είναι μεγάλο και το κόστος στην υγεία. Και για την αντιμετώπιση, την απομάκρυνσή του είναι μεγάλο το κόστος. Καλύτερα λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα στην πηγή. Δεν ξέρω αν είστε τώρα σε θέση να μου δώσετε στοιχεία. Ίσως μπορούσατε να μας τα δώσετε αργότερα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Ζέμπα. Πάβελ Πόκ. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομος. Θα είμαι σαφής πόσο καιρό θα ανέχεται η Επιτροπή τα παιχνίδια που παίζει με μηχανία για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Κούκοβιτς. Κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε, επειδή ε, ο άνθρακας ε, ε, είναι μια σταθερή πηγή μέχρι το 2050 και είναι ο μόνος φυσικός πόρος, η μόνη πρώτη ύλη που έχουμε στην Ευρώπη και είμαστε απόλυτα αυτάρκης, θα ήθελα λοιπόν να στρέψω την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο θέμα αυτό διότι τα εργοστάσια παραγωγής ε, ρεύματος από άνθρακα, με πρώτη ύλη τον άνθρακα, από εκεί ε, προέρχονται πολλές ε, εκπομπές. Από εκεί εκλείεται ο άνθρακας, ο με συγχωρείτε στην ατμόσφαιρα. Οφείλουμε λοιπόν να επενδύσουμε στην έρευνα και επίσης και στην εφαρμογή πιλωτικών προγραμμάτων. Εγώ έχω κατά νου συγκεκριμένου ερευνητέ που ασχολούνται με το θέμα αυτό εδώ και δεκαετίες, όμως αποτελέσματα που να μπορούν να εφαρμοστούν τέτοιου είδου ε, πορίσματα επιστημονικά δεν έχουμε ακόμα. Τώρα λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή για να απαντήσει στις ερωτήσεις που ετέθησαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ε, σημαντικές οι ερωτήσεις που ετέθησαν και ας ξεκινήσουμε με το θέμα του υδράργυρου στα ψάρια. Αυτό δυστυχώς το κληρονομήσαμε από το παρελθόν και δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά σε σχέση με αυτή τη μορφή ρήπανσης. Εκείνο που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι να ελέγχουμε τις χρήσεις ε, υδραργύρου και να υπάρχουν ε, σαφείς κανόνες για το τι είναι επιτρεπτό και τι όχι. Ανεξάρτητα με τις συζητήσεις που γίνονται σε διεθνές επίπεδο, εμείς ασχολούμεται ουσιαστικά με το να ζητήσουμε υποκατάστατα υδραργύρου. Και Δουλεύουμε πάνω σε αυτό ε, προσπαθούμε να περιορίσουμε τη χρήση υδραργύρου στο ελάχιστο. Παραδείγματο χάρη, για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη, με τη στρατηγική που ακολουθούμε για τον υδράργυρο, ε, πλέον δεν υπάρχουν ορυχεία στην Ευρώπη, τα έχουμε αντικαταστήσει και έχουμε και ε, φθήνουσα χρήση υδραργύρου στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για περίπου 200 τόνους το χρόνο για συγκεκριμένες χρήσεις υδραργύρου στην Ευρώπη. Αλλά όπως σας είπα η τάση είναι φθήνουσα. Τώρα για στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο μιλάμε για περίπου 250.000 τόνους σε ετήσια βάση. Και την βιομηχανία στην Ευρώπη. Η ευρύτερη χρήση τερκύρου γίνεται στην χλωροαλκαλική βιομηχανία. Και όλα αυτά υπόκεινται στην οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών. συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών εκπομπών. Η αλήθεια είναι στην ε, χλωροαλκαλική βιομηχανία η τεχνική Mercury Cell δεν θεωρείται ότι είναι και η καλύτερη. Γι' αυτό λοιπόν αναζητούνται αυτή τη στιγμή υποκατάστατα αυτής. Αυτή τη στιγμή η χλωροαλκαλική βιομηχανία στην Ευρώπη έχει έχει τη δική της τη βιομηχανία για να αναζητήσει υποκατάστατα αυτών των κυψελών. Εκτός αυτού υπάρχουν και πολύ περιορισμένες και μικρές χρήσεις του υδραργύρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε μια χρήση στα αμαλγάματα της οδοντιατρικής. Είναι αλήθεια ότι εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει διαμάχη ανάμεσα ε, υπάρχει διάσταση απόψεων όσον αφορά τα οδοντικά αμαλγάματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να διεξάγει μια ανεξάρτητη μελέτη για να αναλύσει ε, τις περιβαλλοντικές πτυχές ε, του θέματος ε, σε σχέση πάντα με τα δοντικά αμαλγάματα και επίκειται η ολοκλήρωση της ε, έρευνας. Βέβαια το θέμα είναι επίκαιρο, γιατί την επόμενη εβδομάδα, 26 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει μία συνάντηση ε, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας περί αμαλγαμάτων. Στην ιστοσελίδα λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το θέμα του υδραργύρου, εκεί ήδη μπορείτε να βρείτε την πρώτη εκδοχή ε, των ε, ερευνητών αυτής της μελέτης. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι ο ΠΟΗ αυτή τη στιγμή προτείνει την σταδιακή μειούμενη χρήση αμαλγαμάτων, όχι όμως την πλήρη κατάργησή της αυτής της χρήσης. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει και άμεση σχέση με το κατά πόσον τα ε, υποκατάστατα που θα αναζητούν θα είναι εξίσου προσιτά ή όχι. Το θέμα του κόστους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των ε, εργοστασίων ε, παραγωγής ρεύματος ή ενέργειας από με άνθρακα, πράγματι είναι αλήθεια ότι αυτά υπάγονται στην οδηγία Περιβιομηχανικών εκπομπών, ε, προβλέπονται ανώτατα όρια εκπομπών, είναι και γνωστές οι τεχνικές ε, και τα φίλτρα που πρέπει να ελέγχονται. Όλα αυτά λοιπόν ε, ελέγχονται από την αντίστοιχη οδηγία και είναι νομίζω σκόπιμο όλα αυτά να συνεχίσουν να ελέγχονται και τα όρια, τα τα όρια να είναι χαμηλά, όσο το δυνατόν πιο χαμηλά γίνεται. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Τώρα, αν μας δοθούν περισσότερα στοιχεία για την παγκόσμια χρήση υδραργύρου σε αιτήσια βάση, τα στοιχεία αυτά θα τα στείλουμε στη Γραμματεία για να σας τα διαβιβάσει περαιτέρω. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, και ευχαριστούμε επίσης ε, και που μας δώσετε μια πολύ καλή εικόνα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις σε διεθνές επίπεδο, γιατί κάποια στιγμή θα κληθούμε και εμείς ως νομοθέτες να τοποθετηθούμε. Άρα δηλαδή φαντάζομαι ε, σύντομα θα ξανασυναντηθούμε. Πάει λοιπόν και αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και προχωράμε τώρα με το υπαριθμόν 20 λέει ο πρόεδρος, προφανώς είναι το 21. Mm -hmm. And, uh, Nos, tisztelt kollégák, elnök úr engem bízott meg, hogy Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Χρότε με παρακάλεσε να τον αντικαταστήσω του Προέδρου, δεδομένου ότι έχει κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις και περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το υπαριθμό 21, μηχανισμός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την κλιματική αλλαγή. το τίτλος. Φαντάζομαι ότι και το αντικείμενο πάντα επίκαιρο για την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Παρακαλώ λοιπόν τον κύριο Ακχάουτ να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όντως, μακροσκελάστατος ο τίτλος αυτής της εκθέσεως. Αλλά μας συμβαίνει συχνά όταν ε, έχουμε νομοθετικά ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την υποπτία ε, και την νομοθεσία περί εποπτείας στον τομέα των αερίων θερμοκηπίου με στόχο να αντικατασταθεί η απόφαση του 2004. 90% των προτινόμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη νέα αυτή πρόταση κανονισμού αντικαθιστά τον παλαιότερο δηλαδή. Ωστόσο ήταν αναγκαία η ε, ενημέρωση των κειμένων για να, δούμε τις, να λάβουμε υπόψη και τις εξελίξεις. Δεν είναι τόσο περίπλοκα λοιπόν τα θέματα, έχουν να κάνουν με την επιτήρηση, με την εποπτεία, αλλά είναι πολύ σημαντικά διότι το αποτέλεσμα πρέπει να είναι η δυνατότητα ε, συλλογής όλων των στοιχείων, να γνωρίζουμε όλα τα δεδομένα, να βλέπουμε αν ε, συνάδουν και με τις συμφωνίες του 2008 και σχέση με τις διεθνείς μας δεσμεύσεις, θα πρέπει και τα κράτη-μέλη στο σύνολό τους να συλλέγουν και να διαθέτουν τα ίδια δεδομένα. Αυτό είναι ο λόγος της ενημέρωσης της νομοθεσίας, της ανανέωσης νομοθεσία, και εμείς ως νομοθέτης ε, καλούμεθα να τοποθετηθούμε επί του κανονισμού για να τον εγκρίνουμε. Όπω έχει λοιπόν η κατάσταση... Η Επιτροπή θα μας εξηγήσει φαντάζομαι σε λίγο, αλλά μπορώ ίσως να σας την προλάβω. Η αναθεώρηση αυτή στόχο έχει να στηρίξει τα κράτη-μέλη στην ε, εφαρμογή του πακέτου μέτρων για, την, ε, για το κλίμα και την ενέργεια. Έχει στόχο να βελτιώσει ταχύτητα διαφάνεια συγκρισιμότητα των δεδομένων. Επίσης, να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη συμμορφώνονται με τις του υποχρεώσεις ω προς την ε, υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση βέβαια, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν την ενίσχυση που δίνεται στι αναπτυσσόμενε χώρε και να παρακολουθεί επίση τη διευκόλυνση ανάπτυξη νέων μηχανισμών αντιμετώπιση τη κλιματική μεταβολή. Αυτή είναι η κύριη στόχη λοιπόν. Ω εισηγητή, συντάσσομαι πλήρω με του στόχου αλλά και με τι προτινόμενε βελτιώσει και θα δείτε ω εκ τούτου ότι στο διατάφτα υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ συγητής, αλλά ελπίζω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντως, κάθε συγητής προτιμά να καταθέτει και κάποιες προτάσεις αλλαγής, τροπολογίες, ελπίζοντας ότι βελτιώνουν το κείμενο και ελπίζοντας ότι θα με στηρίξετε στις τροπολογίες μου, θα ήθελα να σας τις εξηγήσω. Προτείνω λοιπόν την ενίσχυση της πρώτης επιτροπής ορισμένων τομεί. Πρώτον, εκεί όπου γίνεται λόγος για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για το κλίμα, προτείνω να ενισχυθεί και η έννοια περί εκθέσεων ή λογοδοσίας, δηλαδή να περιλάβουμε και τις ρανεώσιμες και το μεριδιό τους στην ε, ενέργεια και άρα επεκτείνω το πεδίο εφαρμογή των διατάξεων περί παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων, ώστε να καλύπτεται και το μερίδιο ενέργεια που προέρχεται από τι ανανεώσιμε πηγέ και την ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργεια. Δεύτερο. δεύτερη πρόταση. Αφού πλέον οι συμφωνίε Κανκούν ορίζουν ότι οι ανεπτυγμένε χώρε οφείλουν να εκπονήσουν στρατηγικέ ή ε, σχέδια ανάπτυξη με χαμηλέ εκπομπέ πέραν του 2020, διατυπώνω την πρόταση στρατηγικές που υποχρεωτικά δυνάμει ε, των συμφωνίων του Κανκούν ε, θα εκπονούν τα κράτη-μέλη. Προτείνω λοιπόν αυτές τις στρατηγικές να συνάδουν με μια οικονομική αποδοτική πορεία προς το μακροπρόθεσμο στόχο για το κλίμα που ορίζεται στο χάρτη πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών. Πρέπει και αυτό να ενταχθεί δηλαδή στην υποχρέωση για ε, υποβολή εκθέσεων για λόγοδοσία από πλευρά των κρατών μελών. Ο μακροπρόθεσμος στόχος. Και τρίτον, σημαντικό πεδίο διεύρυνσης ε, των διατάξεων είναι οι θαλάσσιες μεταφορές, που γνωρίζουμε ότι επίση θα μας απασχολήσουν περαιτέρω στο εγγύ μέλλον και στόχο, έχω να, στόχο έχοντας να διευκολύνω το ε, ζήτημα της συνεργασίας στους στόχους μείωσης των εκπομπών. Προτείνω κάποιες άλλαγες για την νομοθεσία, για τον κανονισμό δηλαδή, ώστε να βελτιωθεί αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών από τα κράτη-μέλη και για τις θαλάσσιες μεταφορές. Αυτές είναι οι κύριες προτάσεις, οι κύριοι στόχοι. Θα δείτε βεβαίως και κάποιες άλλες λεπτομέρειες στις τροπολογίες μου, αλλά αυτοί είναι οι τρεις κύριοι στόχοι. Αυτά είναι τα τρία πεδία στα οποία επιδιώκω να βελτιώσω την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και επίσης, για να καταλήξω, σημαντικό θα είναι το τι θα κάνουμε με τα ε, έσοδα από το σύστημα των ανταλλαγών, το ETS που υιοθετήσαμε το 2008, γιατί αναφέρεται εκεί ότι τουλάχιστον το 50% των εσόδων αυτών θα αξιοποιούνται για τεχνολογία χαμηλής άνθρακα και για τη μετάβαση σε αυτήν. Έτσι λοιπόν σκοπεύω να φροντίσω και στον κανονισμό αυτόν να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, η όρος διαφάνειας για την ε, ικανοποίηση από πλευρά των κρατών μελών του όρου αυτού Τη διάθεση του 50% στην μετάβαση στον, ε, σε οικονομία χαμηλού, χαμηλής περιεκτικότητας άνθρακα. Αυτά είχα να πω εγώ. Περιμένω να ακούσω βεβαίως απόψεις των συναδέλφων, σχεδόν εισηγητών και λοιπόν ε, συναδέλφων της Επιτροπής. Η έκθεση συντάχθηκε σχετικά γρήγορα γιατί είχε ε, χαρακτήρα μάλλον ε, τεχνικό και έτσι προτίμησα να αφήσω περισσότερο χρονικό περιθώριο για τη διατύπωση τροπολογιών ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο και να καταλήξουμε σχετικά γρήγορα στην ε, τελική φάση της διαδικασίας μας. Περιμένω να δω λοιπόν και τις δικές σας αντιδράσεις στην έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Mm. Η Ελίζα Παθηκαρδίνη είναι η πρώτη σκιώδης συγγήτρια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομη. Πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ε, θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι συμφωνούμε για το ποιοι είναι οι στόχοι αυτού του κανονισμού. Είναι λοιπόν αλήθεια, όπως είπε ο συνάδελφος κύριος Άικχουτ, ότι είναι καθοριστική σημασία ο έλεγχος είναι σημαντικό να έχουμε έγκαιρα τα απαραίτητα εντομένα και σωστά στοιχεία σχετικά με τα ε, αέρια θερμοκηπίου. Εξάλλου σημαντικό είναι να βοηθήσουμε και τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή των μέτρων για τη μετώπιση της ε, κλιματικής αλλαγής. Όσον αφορά αυτά τα θέματα όλοι συμφωνούμε. Όμως διαβάζοντας ε, λιγάκι τα θέματα αυτά ε, με περισσότερες λεπτομέρειες νομίζω ότι υπάρχουν κάποια σημεία όπου πρέπει να ε, δώσουμε μεγαλύτερη σημασία να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στη δουλειά που κάνουμε γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να καταλήξουμε σε επικαλύψεις κινδυνεύουμε να καταλήξουμε σε ασάφειες και ασυνέπειες που δεν θα συμβάζονται με άλλους μηχανισμούς ελέγχου. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην φύγουμε από το πλαίσιο αυτής της ε, οδηγίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα λοιπόν να μου επιτρέψετε να σας ε, αναφέρω κάποια στοιχεία, ε, προσκέψη, θέματα τα οποία, επί των οποίων κατά άποψή μου πρέπει να εμβαθύνουμε στις επόμενες εβδομάδες. Παραδείγματο χάρη, όσον αφορά τη στρατηγική ανάπτυξη χαμηλή χαμηλής περιεκτικότητας ε, άνθρακα. Όσον αφορά λοιπόν την υποχρέωση των κρατών μελών να αναπτύξουν συγκεκριμένες προοπτικέ για περιορισμένη περιεκτικότητα άνθρακα και αυτά να γίνουν μέσα σε ένα χρόνο από την έγκριση του κανονισμού, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία κοινοτική νομοθεσία που να προβλέπει τέτοιου είδου υποχρέωση. Έτσι λοιπόν οι αποφάσει που μέχρι τώρα έχουν ληφθεί σε διεθνέ επίπεδο δεν περιλαμβάνουν λεπτομέρειε που να αφορούν στο περιεχόμενο ε, στρατηγικών, που να αφορούν στη δομή, ε, στην χρονική διάρκεια, στο χρονικό πλαίσιο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αναφορά στο χρονισμό, το θέμα του χρόνου. Το θέμα του χρόνου θα αποφασιστεί ε, σε διεθνές επίπεδο, αλλά βέβαια και σε συνδυασμό με άλλα θέματα που ισχύουν. Ε, δεν μπορούμε να εργαζόμεθα για το θέμα αυτό απομονωμένοι και μόνοι. Όσον αφορά τις ε, θαλάσσιες εκπομπές και εδώ πιστεύω ότι τα πράγματα είναι λίγο ασαφή. Δεν ε, γίνεται εξέταση των λεπτομεριών. Ας πούμε, υποχρέωση ελέγχου από τον, των εκπομπών από το θαλάσσιο τομέα. Εκεί Μιλάμε απλώς για ενδείξεις και υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε καλύτερα τα θέματα αυτά, που είναι σημαντικά και δεν μπορούν να παραμείνουν έτσι ασαφή ε, κατόπιν όσον αφορά την ενημέρωση για την κλιματική αλλαγή. Νομίζω λοιπόν ότι και εδώ έχουμε μια παρεμφερή κατάσταση. Γιατί διότι οι πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις εθνικές πράξεις προσαρμογής ή μέτρα προσαρμογής αυτά συνεπάγονται ένα βάρος για τα κράτη-μέλη είτε διοικητικό είτε κόστους, το οποίο αυτή τη στιγμή υποτιμάται σε σχέση με τις, ε, από ό,τι προβλέπετε μέχρι ε, τώρα στις μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου. Και σε αυτό πρέπει να εμβαθύνουμε. Το ίδιο ισχύει και για την ε, τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, εδώ αναφέρεται ότι οι πληροφορίες είναι σε αιτήσια βάση, ενώ δεν ισχύει, είναι σε διετή από ό,τι βλέπουμε. Ε, όλα αυτά βέβαια είναι ένα επιπρόσθετο βάρος και διαρωτώ είναι απαραίτητα όλα αυτά. Μήπως τελικά θα επιβαρύνουμε έναν μηχανισμό τη στιγμή που πολλές φορές προσπαθούμε να είμαστε πιο περιοριστικοί. Υπάρχει λοιπόν το τεράστιο πρόβλημα της επικάλυψης. Βλέπουμε στο άρθρο 20 την ε, αναθεώρηση, εκεί προβλέπεται η αναθεώρηση των ε, εθνικών καταλόγων και της εθνικής απογραφής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει να υπάρχει εσωτερική διαδικασία παράλληλη με αυτά τα οποία ισχύουν σε διεθνές επίπεδο. Αναφέρομαι πάντα στην αναθεώρηση των απογραφικών καταλόγων. Ε, εάν τα αποτελέσματα δεν, είναι, δεν συμβαδίζουν, ε, δεν είναι συνεπή, θα προβλέπεται αυτή η διαδικασία. Και κλείνω. Θα ήθελα να πω το εξής. Εκτιμώ την προσπάθεια του εισηγητή ε, να προσφέρει περισσότερα, να τα κάνει καλύτερα. Αλλά διερωτώ με, γιατί να ασχολείται κανείς με την ενεργειακή απόδοση τη στιγμή που υπάρχει οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ίσως μπορούμε όλο αυτό το θέμα να το εντάξουμε εκεί. Δεν πρέπει δηλαδή να ε, αναγκαστικά να ε, θέλουμε άλλο ένα νομοθέτημα το οποίο απλά θα με το προηγούμενο. Ας πούμε στην Ιταλία εμείς προσπαθούμε να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες ε, να περικόψουμε και νομίζω ότι το κάνουν αυτό και όλοι οι άλλοι γιατί εμείς ας πούμε στην Ιταλία σας λέω διαπιστώνουμε μια τεράστια επικάλυψη νομοθετικών διατάξεων και εδώ πρέπει να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο ε, δεν πρέπει να επιβαρύνουμε τη διαδικασία. Εγώ ε, θεωρώ καταρχήν ως τρόπος εργασίας όλο αυτό είναι λανθασμένο. Ε, και εξάλλου δεν θεωρώ ότι και εδώ είναι η κατάλληλη επιτροπή για να καθορίσουμε νέα όρια εκπομπών. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να επιβαρύνουμε περαιτέρω ε, το όλο νομοθέτημα και την όλη διαδικασία και να κληθεί η Επιτροπή να αντικαταστήσει ένα μηχανισμό έτσι ώστε να είναι πιο γρήγορος, πιο αποτελεσματικός. Θα ήθελα όμως να σας υπενθυμίσω ότι ε, το άριστο δεν είναι φίλος του καλού απαραίτητα. Λοιπόν, Σκιώδη των σοσιαλιστών, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα προσπαθούν να υπολογίσουν, να βρουν έναν τρόπο να αξιολογούμε τι ακριβώς γίνεται, να το μετράμε, ούτως ώστε όσοι υπογράφουν συμφωνίες να μπορούμε να ελέγξουμε εάν κάνουν τις αναγκαίες προσπάθειες να τις εφαρμόσουν. Για το θέμα αυτό όμως έχουν υπάρξει πολλές ε, αντικρουόμενες απόψεις. Μεταξύ με πολλών μεγάλων χωρών όπως γνωρίζουμε. Είναι λοιπόν σημαντικό εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσουμε να δράσουμε ως πρότυπο για τη δημιουργία μεθόδων αποτίμησης και μέτρησης των αποτελεσμάτων, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να δείξουμε, να καταδείξουμε τι κάνουμε και να δούμε τι κάνουν και οι άλλοι. Και αυτό θα πειράσει πολύ και τις άλλες χώρες. Αν δείξουμε ότι τα στοιχεία που συλλέγουμε όλοι είναι συγκρίσιμα, ότι συλλέγουμε τα σωστά στοιχεία, ότι είμαστε ανοιχτοί για το πώς και τι μετράμε. Πρέπει πιστεύω να παίξουμε το ρόλο προτύπου. Αυτή λοιπόν η πρόταση νομίζω ότι είναι καλή, η πρόταση του συγητή. Όπως είπε, είναι ιδιαίτερα τεχνικού χαρακτήρα, αλλά είναι πολύ σημαντική. Γιατί αφορά ε, την αξιοπιστία της ε, κλιματικής πολιτικής όσο θαυμάσιες ε, και αν είναι οι αποφάσεις που λαμβάνουμε εμείς ως Κοινοβούλιο και η Ένωση γενικότερα, όσο φιλόδοξες και είναι οι αποφάσεις μας, εάν, μετά δεν είμαστε σε θέση να καταδείξουμε πως επιτυχάνουμε τους στόχους, δεν έχουν μεγάλο νόημα. Είναι λοιπόν τεχνική αλλά πολύ σημαντική έκθεση. Ο Σκιώδης εισηγήτρια θα προσπαθήσουμε να τη συμπληρώσουμε, να συμβάλλουμε στη βελτίωσή της. Αλλά πιστεύω ότι ο εισηγητής μας μέχρι στιγμής έχει επιτελέσει θαυμάσιο έργο, έχει λάβει υπόψη του το θέμα της ανανεώσιμης ενέργειας, γιατί μιλάμε για ενεργειακή πολιτική, ε, που πρέπει οπωσδήποτε να ε, στοιχειοθετείται με στοιχεία, με αριθμούς είναι πολύ σημαντικό να καλύψουμε και τις θαλάσσιες μεταφορές, την εμπορική ναυτιλία. Για να εφαρμόσουμε την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού, του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας και όσον αφορά τις εκπομπές θείου και τα καύσιμα που περιέχουν θείο στις ε, θαλάσσιες μεταφορές. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε σε ισχύ ένα υψηλής ποιότητας σύστημα για να εποπτεύσουμε την εφαρμογή των αποφάσεών μας. Και κάτι που είναι προφανές. Δεν θέλουμε να είναι άσκοπα περίπλοκο το σύστημα αυτό. Πρέπει να έχουμε σαφή διαδικασία ο στόχος μας δεν είναι να κάνουμε τους έξυπνους, να συμπληρώνουμε πολλά έντυπα. Όχι. Αντίθετα, για να παίξουμε τον ρόλο προτύπου πρέπει οι διαδικασίες μας να είναι σαφείς αλλά και απλές για να αυξήσουμε την αξιοπιστία μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρίς Ντέιβις, επόμενος ο ομιλητής και μετά θα υπάρξουν και άλλοι ομιλητές. Συμφωνώ με τους, προ... με τους προηγούμενους. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε ακριβή πληροφόρηση, ότι την εμπιστευόμαστε. Ότι δεν είναι λανθασμένη, ότι δεν έχει γίνει λαθροχειρία. Όλα αυτά είναι ουσιώδη. Αν θέλουμε να έχουμε αξιοπιστία και στις διαπραγματεύσεις και σε παγκόσμιο επίπεδο και μεταξύ των κρατών μελών και για τη λειτουργία του συστήματος ανταλλαγής ποσοτήτων ποσοστώσεων εκπομπών. Υποστηρίζω λοιπόν τις προτάσεις της Επιτροπής. Μόνο μία ερώτηση. Γιατί ανησυχώ κάπως, όπως και η κυρία Γκαρντίνη, για την επικάλυψη και την υπερβολική γραφειοκρατία. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, εάν η Επιτροπή έχει το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας, και αν θέλει να είναι όσο πιο περιορισμένη γίνεται σε σχέση με αυτό, δεν θα έπρεπε οι προτάση της δεν θα έπρεπε να επιτρέπει να ε, γίνονται εκθέσεις για όλα τα στοιχεία που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Γιατί αυτό ανοίγει τον πίθο των Δαναίδων, μπορεί να, οι βουλευτές να προτείνουν οτιδήποτε. Στην τροπολογία 18 για παράδειγμα λέτε ότι θέλουμε πληροφόρηση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φυσικά. Εμείς εδώ τι χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι υπάρχει αλλού διαδικασία. Αλλά εντάξει, αν δεν υπάρχει αλλού, να υποστηρίξω την πρόταση του συγητή. Αλλά ίσως υπάρχει κάποια επικάλυψη εδώ. Τώρα, α περάσουμε στην τροπολογία 20 που εξετάζει εκπομπέ από τις θαλάσσιες μεταφορές. Υπάρχουν στοιχεία για την ε, μέση ταχύτητα μεταξύ λιμανιών, για παράδειγμα, και το βαθμό συμμόρφωσης με διάφορους κανονισμούς. Φυσικά να συμμορφούνται με τους κανονισμούς. Αλλά θα ήθελα να μάθω ποιο θα ε, βρίσκει αυτή την πληροφόρηση. Αυτός είναι ο καλύτερο τρόπο για να την συλλέξουμε αν θέλουμε να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί και όσο λιγότερο γραφειοκρατικοί γίνεται. Και τέλος για την τροπολογία 26, όπου ο εισηγητής θέλει πληροφορίες για το βαθμό στον οποίο η δράση του κράτους μέλους συνάδει με μια οικονομικά αποδοτική πορεία προς το μακροπρόθεσμο στόχο της Ένωσης για το κλίμα. Ε, νομίζω ότι είναι δύσκολο ένα κράτος μέλος να κάνει κάτι τέτοιο πολιτικά θα το έφερνε και σε πολύ δύσκολη θέση. Θα ήταν καλό αν θα μπορούσε. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα ψήφιζα υπέρ ή κατά μια τέτοια τροπολογία. Θα ήθελα τη γνώμη της Επιτροπής για το θέμα αυτό. Καλώς ευχαριστώ. Θα δούμε τι έχει να πει και η Επιτροπή. Όμως έχω ακόμα τρεις συναδέλφους περιμένω να λάβουν το λόγο. Έτερος, για να μην περιορίσω το χρόνο ομιλίας, αλλά θα σημειώσω και τον κύριο Πρόντι και μετά τους άλλους Παρακαλώ, κύριε Πρόντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι αναμφίβολα πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έγγραφο διότι η ε, κλιματική πολιτική βασίζεται σε γεγονότα, πρέπει να βασίζεται σε αδιαμφισβήτητα στοιχεία. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ε, το πόσο σημαντικό και αναπόφευκτο είναι να επικαιροποιούμε τις παρατηρήσεις μας και αναφέρομαι κυρίως ε, στο GMS ε, στον ε, δορυφόρο για το παρακολούθησης για το περιβάλλον και την ασφάλεια. Ε, γιατί με τον τρόπο αυτό ο δορυφόρος αυτός μπορεί να δώσει πάρα πολλές πληροφορίες για το σύνολο του πλανήτη, για το τι ακριβώς συμβαίνει σε θέματα εκπομπών. Πρόκειται λοιπόν για δεδομένα τα οποία είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα, λεπτομερή και αφορούν όλα τα αέρια θερμοκηπίου τα οποία ε, εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ότι η διάταξη των δορυφόρων οι δορυφόροι θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην είναι κάτι που να επαφείται στην καλυτέληση των κρατών μελών. Ε, πρέπει λοιπόν να εντάσσονται οι δορυφόροι ως μια απαραίτητη υποδομή για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο δεδομένων που δείχνουν τη συγκέντρωση ε, αερίων του θερμοκηπίου. Ε, να υπάρχει επίσης ε, και η δυνατότητα ε, να εντοπίζονται οι τροχές των, των αερίων θερμοκηπίου, ακριβώς όπως συμβαίνει και με τον καπνό που βγαίνει από μία καμινάδα. Είναι λοιπόν καθοριστική σημασίας να έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο όταν θα επικαιροποιηθεί θα είναι και λιγότερο βαρύ για τα κράτη-μέλη, γιατί το πλαίσιο αυτό θα αποτελείται από... σε αυτό θα εντάσσονται διάφορα οργανισμοί, γραφεία και θα υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει σύγκριση δεδομένων ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά και γενικότερα σε όλα τα κράτη στον πλανήτη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ζήμπα. Ε, ο κύριος Ζήμπα. Μάλλον μετά ο κύριος Ζήμπα. Ε, κύριος Γκουζή, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να, καλώ, να ευχαριστήσω, κύριος Γκουσί, τον ε, εισηγητή και να διατυπώσω και εγώ από μου την ερώτηση που ακούσαμε από άλλους ομιλητές. Δηλαδή το κατά πόσον συνάδουν, κατά πόσον υπάρχει ε, της χαρακτηριστικών μεταξύ αυτών που πράττουμε στην Ευρώπη και αυτών που μπορούν να γίνουν σε διεθνές επίπεδο. Χωρίς να θέλω να ε, διαφοροποιηθούμε, θέλω απλώς να είμαστε πιο αξιόπιστοι και βέβαια πιο απλοί μια ερώτηση που απευθύνεται δηλαδή στον εισηγητή αλλά και στην Επιτροπή που ασφαλώ θα λάβει το λόγο φαντάζομαι διότι διαγνώσκω ένα πρόβλημα κυριαρχίας. Υπάρχουν κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη είναι συνηθισμένα, δέχονται την ε, εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Έχουμε δηλαδή οργανισμούς όπως η Επιτροπή ε, που δίνουν, λαμβάνουν φάση αλλά και εποπτεύουν τα ε, κράτη-μέλη. υπάρχουν άλλα κράτη, θα έλεγα πιο ανατολικά, τα οποία δεν δέχονται να ελεγχθούν και να αμφισβητηθούν οι δηλώσεις τους από κάποιον που θα τους πει «Α, δεν ήταν αξιόπιστες οι δηλώσεις». Άρα και δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, γι' αυτό λέγω, χρησιμοποιώ τον όρο ανατολικά κράτη, αλλά τα κράτη αυτά τα ανατολικά ε, έχουν μια διαφοροποίηση ως προς την πολιτική πρακτική. Επίσης, μια και έχω επισκεφθεί πολλές ε, τέτοιες διασκέψεις κλιματικού χαρακτήρα, με αντικείμενο το κλίμα. Υπάρχουν διάφορα επιστημονικά δεδομένα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και, το, και τις συνέπειες αυτού στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, ή επιμέρους στα διάφορα κρατημένα κλπ. Υπάρχουν λοιπόν επιμέρους ε, δεδομένα, αλλά ξέρετε ότι όλα αυτά προκύπτουν, με, όπως το γνωρίζουμε όλοι βέβαια, μέσα από ένα παζάρι, μέσα από μια διαπραγμάτευση πολιτικού χαρακτήρα. Δηλαδή έρχονται μεν οι επιστήμονε και δίνουν τα στοιχεία του, αλλά μετά οι υπουργοί και αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων ακόμη ε, συζητούν μεταξύ του και λένε ναι, να υπογράψουμε μια πολιτική δήλωση Φερρυπίν Κοπεχάγη, αλλά να κοιτάξουμε και λίγο και κάποιε τροποποίησει στο Κιώτο πολύ ευχαρίστω, αλλά δώστε μας 150.000 ε, τόνους περιθώριο, όπω είχε συμβεί στην περίπτωση της Ρωσίας, σε παραδείγματι. Ε, μην ξεχνάμε ότι το 90 η κατάσταση δεν ήταν αυτή που γνωρίζουμε σήμερα. Και έτσι, παρά την αυστηρή επιστημονική γνώση που εμείς οφείλουμε να έχουμε, τελικά όλα αυτά καταλήγουν σε ένα πολιτικό παζάρι, το οποίο ξεφεύγει βέβαια από τα ακριβή επιστημονικά στοιχεία. Άρα λοιπόν θα ήθελα να γνωρίζω, δεν ξέρω αν είναι εύκολο, αλλά ίσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θα μα δώσουν κάποιε ενδείξει και ίσως και από πλευρά του Συμβουλίου, αν μπορούμε να πείσουμε τους εταίρους που έχουν ήδη φερειπίν ε, υπογράψει την, ε, το πρωτοκόλλο του Κιώτο. Πολύ ωραία λοιπόν. Ε, προηγουμένως έγινε μια μικρή παρεξήγηση, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά τώρα πραγματικά έχει το λόγο ο κύριος Ζέμπερ. Κοιτάξτε, και εμένα τα ουγγρικά μου δεν είναι και τόσο καλά, για να μπορώ να σας καταλαβαίνω απευθείας. Λυπάμαι και εγώ, δεν κατάλαβα καλά. Η έκθεση λοιπόν που μας ε, παρουσιάστηκε είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη και θα τολμούσα να πω ότι ξεπερνάει κατά πολύ το στόχο μας. Αλλά ε, έτσι κι αλλιώ, εγώ δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από τον εισηγητή ε, με το δυναμισμό που τον χαρακτηρίζει. Νομίζω το ε, καθοριστικό στοιχείο θα πρέπει να είναι ότι προσπαθούμε να συστήσουμε σε διεθνές επίπεδο ένα σύστημα ελέγχου. Δίνω δίκιο στον συνάδελφό μου ότι εμείς στην Ευρώπη θα πρέπει να αποτελούμε παράδειγμα προς μίμηση, αλλά και αυτό μέχρι ενός ορίου. Γιατί κατά την άποψή μου αυτό που παρουσιάζεται σήμερα είναι υπερβολικό. Ε, θα ακούσουμε μετά τι θα πει ο κύριος Μέτσκια από την Κομισιόν αλλά νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλη δυσκολία η Κομισιόν να συμπεριλάβει όλα αυτά και να τα ελέγχει. Και δεύτερον, είναι δύσκολο να ε, εφαρμοστούν όλα αυτά σε επίπεδο κρατών μελών. Γιατί αυτός ο κορσές που μας ε, επιβάλλεται μπαίνει και σε πάρα πολλές λεπτομέρειες και μάλιστα αφορά και τομεί ε, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι εκτός. Αν δούμε λοιπόν τις διάφορες ε, τροπολογίες ε, θα δούμε ότι έχει έναν κατάλογο ε, κυρίως όσον αφορά το νοτικό χάρτη από το 20 μέχρι το 50 όμως είναι διαφορετική η δική μας η θέση. Εμείς μιλάμε για ορόσημα και όχι για στόχους και αυτό έτσι πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση. Τώρα, ό,τι δεν επιτεύχθηκε από την άψη των πρασίνων στην ε, πολιτική για το κλίμα περιλαμβάνεται εδώ. Αυτό όμω είναι λάθος. Αυτή είναι τεχνική η έκθεση και σε τελική ανάλυση αυτό που ενδιαφέρει είναι το δίκαιο που θα ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 20 να εφαρμόζεται σωστά, να υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία για να μπορούμε να πάμε σε διεθνείς διαπραγματεύσεις και να προχωρήσουμε στο θέμα της ε, κλιματικής αλλαγής. Το θέμα δεν είναι τι μας αρέσει και τι επιθυμούμε, γιατί δεν είναι Χριστούγεννα. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να παραμείνουμε ρεαλιστές. Και διαβάζοντα, α πούμε, ότι θα πρέπει να υπάρχουν ιδιωτικέ πηγές χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση κοινωνικής αλλαγής, κάνει η τροπολογία υπερθυμών 4, εδώ κινούμεθα ε, σε κινούμενη άμμο. Ε, και πάρα πολλά. Αυτά που λέγονται για το LULUCF, παραδείγματο χάρη. Εδώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τη χρήση γης, αλλαγή στη χρήση γης και ε, δασοκομικές δραστηριότητε. Επίσης και για τις θαλάσσιες εκπομπέ και εκεί να είμαστε προσεκτικοί. Νομίζω ότι ως κοινότητα ακόμα δεν έχουμε οριστική και αμετάκλητη άποψη. Ε, εντάξει, αυτέ τι τροπολογίε, εμεί θα τι δούμε ω ομάδα και θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε μια ρεαλιστική χρειά. Και συγγνώμη κιόλας, ε, δεν μπορώ να περιμένω την ε, ε, απάντηση Κομισιόν, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα υδάτων. Σε λίγο θα μιλήσει ο επίδρομος κ επίτροπο ε, αρμόδιο του περιβάλλοντο και γι' αυτό παρακαλώ να γράψει τα πρακτικά με όλε τι λεπτομέρειε αυτά που θα λεχθούν από τώρα και μέχρι το τέλο τη Επιτροπή για να μπορώ να τα διαβάσω. Δεν έχει δει κανεί άλλο το λόγο, αλλά επαναλαμβάνω, μήπω θέλει κανεί άλλο το λόγο. Όχι. Έγιναν πολλές ερωτήσεις προς τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κύριος Δευτής θα μας απαντήσει. Ευχαριστώ που μας καλέσατε και μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ την Επιτροπή. Νομίζω ότι όλοι όσοι μίλησαν υποστήριξαν σε μεγάλο βαθμό την πρόταση της Επιτροπής. Να ξεκινήσω λοιπόν όπως και ο συγητής, λέγοντας ότι δεν είναι κάτι το εντελώς καινούριο. Πρόκειται για εποπτεία και <clears throat> υποβολή εκθέσεων για το θέμα αυτό. Αυτό το κάνω από το 1992. Έχουμε λοιπόν ε, πολύ πείρα για το πώς ε, να επιτηρούμε και από καιρούς καιρό βελτιώνουμε το σύστημα εποπτείας. Το κάναμε όταν ε, εγκρίθηκε η Συμφωνία του Κιώτο και τώρα είναι δεύτερη φορά γιατί περνάμε σε νέα φάση με το 2013 Εγκρίναμε Ευρωπαϊκή Νομοθεσία το πακέτο κλίματος και ενέργειας, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν σε κάποια άρθρα τροποποιήσεις. Δεύτερον, σε διεθνές επίπεδο, συμφωνήσαμε να βελτιωθεί ο έλεγχος, η επαλήθευση και η υποβολή εκθέσεων. Έγινε μεγάλη συζήτηση μετά τη συνάντηση το Παλί το 2007. Κατέληξαν οι συζητήσει αυτές στο Durban πέρυσι και ήδη προηγουμένως στο Κανκούν. Οπότε χρειάζονται κάποιες αλλαγές στην νομοθεσία. Και τρίτον, έχουμε και τη στρατηγική Ευρώπη 2020 με τους κύριους στόχους και την ανάγκη υποβολής εκθέσεων που πρέπει λοιπόν οι στόχοι αυτοί να μεταγραφούν σε νομοθεσία. Έχουμε υπόψη μας ιδιαίτερος από πλευράς Επιτροπής ότι πρέπει στα κράτη-μέλη να τους επιφορτίζουμε με υπερβολικά καθήκοντα όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων. Έχουμε κάνει λοιπόν μια αναλυτική μελέτη επιπτώσεων για να δούμε τι κόστος έχουν οι τροποποιήσεις που θέλουμε να εφαρμόσουμε και δεν νομίζουμε ότι είναι υπερβολικό αυτό το επιπλέον κόστος. Μπορούν να το φέρουν τα κράτη-μέλη, κατά τη γνώμη μας, γιατί Πολλές από τις υποδομές είναι ήδη, λειτουργούν ήδη και για μια σειρά αποζητήματα, αλλά υπάρχει ήδη υποδομή. Τώρα, για παράδειγμα, πρέπει να μας υποβάλουν εκθέσεις για την οικονομική βοήθεια προς τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Τις εκθέσεις αυτές τις κάνουν ήδη προς τον ΩΣΑ. Τώρα θα πρέπει να τις αποστέλουν σε εμά και σε εμάς γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τμήμα του UNCCC και του πρωτοκόλλου του Κιώτο, άρα πρέπει και εμείς να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που έχουμε. Έχουμε τέτοιες υποχρεώσεις σε διεθνές επίπεδο. Και περί αυτού πρόκειται κυρίως αυτή την νομοθεσία, να μας επιτρέψει να υποβάλουμε τις εκθέσεις που πρέπει σε διεθνές επίπεδο. Έχουμε κατά νου ότι πρέπει να αποφεύγουμε λοιπόν τις επικαλύψεις. Γι' αυτό λοιπόν στους μηχανισμούς επιτήρησης δεν θα δείτε καμία αναφορά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποδοτικότητα της ενέργειας γιατί αυτά τα θέματα τα ρυθμίζουμε αλλού. Δεύτερον, συγκεκριμένη ερώτηση για τις θαλάσσιες μεταφορές. Συνεχίζονται οι συζητήσεις και εντός των υπηρεσιών μας. Εκτελούνται οι μελέτες επιπτώσεων για να δούμε ποιος θα ήταν ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και αυτό αφορά και τις ανάγκες επιτήρησης. Σε αυτό το νομοθέτημα απλώς λέμε ότι κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να γίνεται κάποια, να υποβάλλονται κάποια στοιχεία για τι μεταφορές, αλλά αργότερα θα καθορίσουμε πια μέσω πρωτογενού νομοθεσίες που θα πρέπει να αποφασίζει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Τι δηλαδή ακριβώ θα περιέχουν αυτές οι εκθέσεις. Πολλές λεπτομέρειες για τα ακριβή στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται. Στο παρελθόν τις ρύθμιζαν κατ' εξουσιοδότηση πράξης. Είχαμε την απόφαση για την εφαρμογή του ε, μηχανισμού παρακολούθησης. Τώρα προστίθεται το νέο νομοθέτημα. Σε διεθνές επίπεδο τόσο λεπτομερή ε, στοιχεία δεν υπάρχουν. Γι' αυτό αυτές οι λεπτομέρειες θα τι αναφέρουμε στην περαιτέρω λεπτομεριακή νομοθεσία. Αλλά έχουμε δεσμευθεί διεθνώς να κάνουμε εκθέσεις για τις ε, χρηματοοικονομικές ροές και τι υποστήριξη δίνουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τι ακριβώς θα περιέχουν οι εκθέσεις θα το δούμε αργότερα. Και θα αναφερθεί αργότερα σε κατεξουσιοδότηση πράξη. Αλλά χρειαζόμαστε να έχουμε αυτή τη γενική αναφορά. Για ένα χρόνο θα έπρεπε να επανέλθουμε και να ζητήσουμε άλλη μια τροποποίηση στον ε, κανονισμό για την ε, παρακολούθηση. Τέλος. για το θέμα των ακρογωνιαίων λίθων συγγνώμη, μάλλον, μάλλον των όροσίμων. Συζητιούνται αυτή τη στιγμή με το Συμβούλιο. Έχει υπάρξει μόνο μία ανακοίνωση της Επιτροπής που αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά δεν έχει υπάρξει απόφαση του Συμβουλίου, οπότε σε αυτό το νομοθέτημα, στο οποίο μιλάμε για τις εκθέσεις, δεν κάνουμε καμία αναφορά στο θέμα των οροσίμων γιατί δεν έχει ακόμη αποφασιστεί. Ξέρετε ότι μιλάμε για αιτήσει εκθέσεις τώρα. Όταν κατόπιν θα θέλουμε να κάνουμε πιο, πιο λεπτομερή επιτήρηση και το εάν τηρούμε το πρόγραμμά μας, τότε θα κοιτάξουμε το πακέτο ενέργειας και διεθνώς τι θα κάνουμε για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης για το Κιώτο μέχρι το 2020 και για τα θέματα αυτά ήδη στην νομοθεσία υπάρχουν απαιτήσει προς τα κράτη-μέλη να κάνουν προβλέψεις και προβλέπουμε να γίνονται σε αιτήσια για να βλέπουμε κατά πόσον τηρούμε αυτά που έχουμε αποφασίσει και για να δώσουμε και τις αναγκαίες συστάσεις στα κράτη-μέλη αν χρειάζεται. για την ερώτηση όσον αφορά την επανεξέταση των εθνικών μητρών. Είναι αρκετά περίπλοκο το θέμα αυτό. Έχουμε την έννοια της ε, ε, διακρύβωσης ποιότητας, κάτι που μας ζητείτε διεθνώς. Πρέπει να κάνουμε έναν εσωτερικό έλεγχο ποιότητας. Έχουμε την υποχρέωση αυτή. Και υπάρχει και μία διεθνής επανεξέταση που προβλέπεται από το UNCCC. Δεν την αντικαθιστούμε λοιπόν. Ούτε επικαλύπτουμε, ούτε κάνουμε δύο φορές τη δουλειά. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε ότι τα στοιχεία που δίνουμε στη διεθνή επανεξέταση έχουν ελεγχθεί ως προς την ποιότητά τους. Πρόκειται λοιπόν για συντονισμένη δράση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για το Περιβάλλον και της Εθνικές Διοικήσεις είναι απόλυτα αναγκαίο. Είναι διεθνής υποχρέωσή μας. Διεθνής υποχρέωσή μας. Νομίζω ότι απάντησα σε όλα όσα υπόθηκαν που σχετίζονται με την απόφαση για τον μηχανισμό παρακολούθησης. Δύο ερωτήσεις ε, πήγαιναν παραπέρα. Η ερώτηση του κ. Πρόντι και η πρότασή του για το σφαιρικό σύστημα παρακολούθησης της ε, περιβαλλοντικής ασφάλειας. Βεβαίω το υποστηρίζει ιδιαίτερο Κομισιόν αυτών. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος ε, παρακολούθησης, όχι από κάτω προς τα πάνω, αλλά από κάτω τα πάνω, από πάνω προς τα κάτω, συγγνώμη. Αλλά δεν έχει συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο, στα πλαίσια του UNCCC, αλλά θα μπορούσε να μας παράσχει συμπληρωματική πληροφόρηση και γι' αυτό τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή αποφάσισαν να βαδίσουν και αυτή την οδό. Αλλά είναι εκτός της εντολής του συγκεκριμένου νομοθετήματος. Και τέλος, το θέμα αυτό μεταφοράς κυριαρχίες. Το κείμενο που σας προτείνουμε δεν ζητάει καμία μεταφορά κυριαρχίας από τα κράτη-μέλη προς την Ένωση. Το μόνο που ζητάμε είναι τα κράτη-μέλη να μας υποβάλουν εκθέσεις. Αυτό δεν είναι μεταφορά κυριαρχίας. Τα θέματα κυριαρχίας τίθενται πάντα όσον αφορά την έκθεση, τι στοιχεία δηλαδή θα μας στείλετε, τι επίπεδο, διασφα... Ε, τι επίπεδο διαφάνειας πρέπει να διασφαλίζετε. Αλλά αυτά που προτείνουμε εδώ για το επίπεδο διαφάνειας που πρέπει να έχουν τα στοιχεία έχει, έχουν ήδη συμφωνηθεί σε διεθνή φόρα και σε άλλα νομοθετήματα της Ένωσης. Αυτό λοιπόν το νομοθέτημα προσπαθεί να διασφαλίσει ότι θα έχουμε την παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση που χρειαζόμαστε για να ελέγχουμε την εφαρμογή της υπαρχούσης νομοθεσίας. και προσβλέπω στη συζήτηση για το θέμα αυτό της προσεχής εβδομάδας και ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα γιατί την πρώτη πρώτη του 13 θα πρέπει να τα εφαρμόσουμε και δεν απέχει και τόσο πολύ. Σας ε, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Διευθυντά για αυτές τις απαντήσεις που μας δώσετε. Ε, ακόμα ένας συνάδελφος ε, έχει ζητήσει τον ε, λόγο ε, συγκεκριμένα ο εισηγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους τους ε, σκιώδεις για τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε πολύ και για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Αυτό που έμαθα είναι ότι μπορεί κανείς να είναι και υπερβολικά δυναμικός. Ε, δεν ξέρω, ε, εγώ θέλω να το κλάβω σε κοπλιμέντο αυτό που μου έκανε ο κύριος ε, Ζίμπερ και τον ευχαριστώ πολύ για το, γιατί σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομίζω ότι πρέπει να είμαστε δυναμικοί. Εγώ ε, με μεγάλη μου χαρά ε, θα περιμένω τους ε, συμβασμούς, αποκοινούμε τους σκιώδης ηγητές. Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως κράτη-μέλη έχουμε δεσμευτεί για τα προγράμματα περιορισμένης χρήσης του άνθρακα. Στο Κανκούν το κάναμε αυτό. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να μας στείλετε πληροφορίε, για το πώ αυτό μπορεί να γίνει αποτελεσματικά από πλευρά κόστους. Αυτό ε, είναι λογικό και δεν έχει σχέση ούτε με δυναμισμό ούτε με τίποτα. Ε, με την οικονομία έχει σχέση, με απλά οικονομικά. Άρα δηλαδή όταν κοιτάμε λίγο τον χάρτη πορείας κομισιών για ε, περισμένη χρήση για, μάλλον για περισμένες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αυτό που με εκπλήσει, αν άκουσα καλά αυτά που είπε ο κύριος Ζέμπερ, ακόμα και το να το πει κανείς, ε, του φαίνεται υπερβολικό. Όσον αφορά τώρα την ε, έκταση των ανωμένων πηγών ενέργειας και την αποτελεσματικότητα. Κανείς μας δεν θέλει να επιβαρύνει πολύ την ε, γραφειοκρατία. Αλλά όπως υπόθηκε και προηγουμένως, αν δούμε την ε, μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου, δεν είναι φοβερή η γραφειοκρατία. Απλά αυτά είναι δεδομένα που υπάρχουν έτσι κι Το σημαντικό είναι ότι οι πληροφορίες <coughs> υπάρχουν, αλλά δεν είναι αρμονισμένες και αυτή είναι η μόνη κατάλληλη στιγμή που μπορούμε να επιτύχουμε, να επιβάλλουμε την αρμόνιση μέσα από νομοθετικές πράξεις. Άκουσα τον συνάδελφο ε, ίσως να μην το αρέσουν αυτά που ελέγχθησαν που έχουν σχέση και με άλλες γενικές διευθύνσεις. Αλλά υπάρχουν οι πληροφορίες. Ε, δέστε λιγάκι την Eurostat. Υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Τις δίνουν τα κράτη-μέλη, όχι όμως ε, εναρμονισμένα, με εναρμονισμένη διαδικασία. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν την νομοθεσία για να το πετύχουμε. Τώρα, όσον αφορά τα σκάφη, την ναυτιλία, ε, κοιτάξτε, Υπάρχουν ε, πάρα πολλές επιστημονικές ε, μελέτες ε, που δίνουν έτσι κάποια γνώση, δίνουν πληροφορίες για τους δείκτες και οι επιστήμονες μου λένε ότι αυτό είναι καθοριστική σημασία. Εγώ λοιπόν είμαι ανοιχτός ε, και για άλλους δείκτες, αλλά αυτοί οι δείκτες είναι απαραίτητοι για να ασχοληθούμε και με την, ε, ε, τις θαλάσσιες μεταφορές. Και ο στόχος, που δεν είναι, βέβαια, να καθυστερήσουν πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε τελική ανάλυση εδώ πρόκειται για νομοθετικές νομοθεσία που αντικαθιστά την ήδη υπάρχουσα, όπως είπε ο Άρθουρ. Εδώ και 20 περίπου χρόνια κάνουμε ελέγχου. Τώρα πλέον δεν απεμπολούμε κυριαρχικά δικαιώματα, απλά ενημερώνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με εναρμονισμένο τρόπο έτσι ώστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να ανταποκριθεί στις ε, ε, υποχρεώσεις που αναλαμβάνει σε διεθνές επίπεδο. Κάνει για τέλη επιπρόσθετο βάρος, όμως θέλουμε εναρμόνιση για να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιόπιστος εταίρος και χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στοιχεία και για μελλοντικέ πολιτικές, όπως είναι οι θαλάσσιες μεταφορές. Άκουσα ερωτήματα από τον Κρίς, άκουσα και την υποστήριξη που εξέφρασε η συνάδελφος Εκείνο που ενδιαφέρει είναι σε τελική ανάλυση είναι το Κοινοβούλιο να έχει ισχυρή θέση, να υπάρχει το σωστό μείγμα καλών εναρμονισμένων πληροφοριών, χωρί υπερβολική γραφειοκρατία, παράλληλα όμω και πληροφορίε, οι οποίε μακροπρόθεσμα θα μας ε, επιτρέψουν να εφαρμόσουμε στρατηγικές περιορισμένων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, παράλληλα όμω με σχεση κόστου κόστους-οφέλους. Δέστε λοιπόν λιγάκι τη συμφωνία του Κανκούν. Εκείνο που προσπαθώ να κάνω είναι ε, όλα αυτά να γίνουν, όπως σας είπα, με εναρμονισμένο ε, τρόπο, ε, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους-οφέλους. Σαν αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η πρώτη φορά που εμείς ως Κοινοβούλιο ζητάμε από την Επιτροπή να είναι λίγο περισσότερο φιλόδοξη, ε, να ανοίξει τη συζήτηση και με άλλες γενικές διευθύνσεις. Αλλά εν πάση δώσει, τώρα δεν είναι δική μας υπόθεση αυτό να το ε, ζητάμε. Ε, για μας αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε σωστές πολιτικές. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ συνάδελφοι και εγώ. Και εύχομαι επικοδομητική δουλειά στην έκθεση αυτή. Για να είναι όμως επικοδομητική, σας υπενθυμίζω τις προθεσμίες για την κατάθεση τροπολογιών. 28 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι, η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας προβλέπεται για τις 30 Μαΐου και κατά πάσα πιθανότητα στην Ολομέλεια του Ιουλίου, πριν ακριβώς από τις τελευταίες διακοπές δηλαδή, θα έχουμε την ευκαιρία να εγκρίνουμε την έκθεση στην ε, Ολομέλεια. Μια ακόμη ε, πληροφορία, προσεχής μας συνεδρίαση είναι η 25η Απριλίου και η επόμενη 26, 25 και 26 Απριλίου, δηλαδή μετά τις διακοπές του Πάσχα και μέχρι τότε σας εύχομαι καλή δουλειά και καλή ξεκούραση.